Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Και επιτρέψτε μου να κηρύξω την έναρξη της συνεδρίασής μας της Υποπιτροπής για την Ασφάλεια και Άμυνα. Πρώτα απ' όλα, πρώτη μου ανακοίνωση αφορά την διερμηνία και τις γλώσσες που είχαν προτεραιότητα ε, σήμερα και που είναι βέβαια οι γλώσσες των τακτικών μελών της υποπιτροπή μα. Επίσης πρέπει να ξέρετε όταν μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας. Και τώρα θα ήθελα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη παρακαλώ. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις θεωρώ ότι εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Ανακοινώσεις της Πρόεδρου τώρα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη εκμαρουσμού και της γραμματείας για το χάος που δημιουργήθηκε λίγο με τη σημερινή συνεδρίαση που αποφασίσαμε να αρχίσει αργότερα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το βραβείο Σαχάροφ. Οπότε τα μέλη της Επιτροπής μας, ακόμα και πολλά αναπληρωματικά, συμμετέχουν και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, την ΑΦΕΤ. Γι' αυτό. Συνεπώς, ας περάσουμε στην ημερήσια διάταξη τώρα αυτή καθεαυτή. Το πρώτο σημείο, που είναι η δεύτερη εξέταση της έκθεσης για τις εξαγωγές όπλων. Εφαρμογή της κοινή θέσης 2008 κάθετος 944. Η συγκίτρια μάλλον, είναι η κυρία Βαλέρο. Έχουμε και τους σκιώδεις εισηγητές. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ήταν 23η Σεπτεμβρίου, αν δεν απατάει η μνήμη μου. Γνωρίζω ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα σχετικά με την συνεδρία των σκιωδών εισηγητών. Οπότε θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Μποντήλ Βαλέρο πρώτα απ' όλα να μας εξηγήσει την κατάσταση. Στην επόμενη συνεδρίασή μας, στις 12 Νοεμβρίου, πάλι θα έχουμε λίγο χρόνο, γιατί στις 16 Νοεμβρίου τελικά θα ψηφίσουμε, οπότε υπάρχει λίγος χρόνος ακόμα για λιγμούς. Ας ακούσουμε όμως την κυρία Βαλέρο να μας εξηγήσει την κατάσταση. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τις 180 τροπολογίες που υποβλήθηκαν και που πιστεύω ότι θα ε, συμβάλλουν σε ένα καλύτερο τελικό αποτέλεσμα. Επίσης πιστεύω ότι παρότι οι τροπολογίες αυτές ε, αντιπροσωπεύουν ένα πολύ ευρύ φάσμα απόψεων, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό ε, που να μπορεί να γίνει αποδεκτός από όλους. Όταν ξεκινήσαμε τις εργασίες πάνω στο θέμα αυτό, η σκέψη μου ήταν ότι όσον αφορά την κατάσταση ασφαλείας στις περιοχές της γειτονίας μας έχει αλλάξει η κατάσταση και ότι Τώρα υπάρχουν πιο σημαντικές απαιτήσει απέναντι στους ε, ευρωβουλευτές. Ε, θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά την κατάσταση. Και περισσότερο από ό,τι πιθανότατα χρειαζόταν στο παρελθόν, θα πρέπει να φροντίσουμε τα όπλα να μην καταλήγουν σε λάθος χέρια. Επίσης, επέλεξα να επικεντρωθώ στον ρόλο του Κοινοβουλίου, αλλά και στην διαφάνεια όχι μόνο για το Κοινοβούλιο, αλλά και για το κοινό. Είμαστε υπεύθυνοι, έχουμε μια ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Ε, θα πρέπει να γνωρίζουν πώς ε, πραγματοποιούμε τις ε, κοινοβουλευτικές μας εργασίες. Έχουμε λοιπόν τη νέα κατάσταση ως προς την ασφάλεια και από την έκθεση Co-Arms μπορούμε να μάθουμε σχετικά με τα λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν έγιναν όλα σωστά. Κάνουμε και εμείς λάθη, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε τους κανόνες που υπάρχουν. Υπάρχουν διάφοροι κανόνες, υπάρχουν και διάφορες απόψεις για τους κανόνες αυτούς και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε λύση. Υπάρχουν μερικοί που πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει ενιαία ερμηνεία ότι όλοι θα πρέπει να εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες, ε, ενώ άλλοι δεν πιστεύουν ότι οι χώρες που έχουν προχωρήσει πιο πολύ θα πρέπει να μειώσουν το επίπεδο ασφαλείας τους. Ε, κάτι τέτοιο άλλωστε ε, θα ήταν εις βάρος της αξιοπιστίας μας. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία λύση με την οποία να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Η κοινή προσέγγιση είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις που έχουμε, αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε αυτό και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν πιο αυστηρούς κανόνες εφόσον το θέλουν. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να μπορούμε να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό που ανέφερα στην εισαγωγή μου. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν. Και βέβαια εύκολο είναι να κάνει κανείς τον έξυπνο εκ των υστέρων, αλλά ίσως θα έπρεπε να έχουμε αξιολογήσει καλύτερα την κατάσταση στις χώρες προς τις οποίες πουλήσαμε όπλα. Ελπίζω λοιπόν στην έκθεση να μπορέσουμε να το συμπεριλάβουμε και αυτό. Να πρέπει όχι μόνο να κοιτάμε το υλικό αυτό καθεαυτό, όχι μόνο δηλαδή τι όπλο στέλνουμε σε ποια χώρα και σε ποιον τελικό χρήστη, θα πρέπει να εξετάσουμε και την κατάσταση γενικά στη χώρα και στην περιφέρεια. Και να μην επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στο υλικό που εξάγουμε. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις και σε αυτά τα θέματα. Μία ερώτηση σημαντική όπου έχουμε διαφορετικές απόψεις έχει να κάνει με τους τελικούς χρήστες. να μην καταλήγουν τα όπλα σε άλλους χρήστες τελικά από αυτούς που θεωρούμε εμείς τελικούς χρήστες. Και εδώ δεν αρκούν τα πιστοποιητικά. Θα πρέπει εμείς να ελέγχουμε καλύτερα εκ των υστέρων την κατάσταση. Αυτό μπορεί να στοιχήσει ε, κάτι παραπάνω για τα κράτη-μέλη, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και να βρούμε ένα μοντέλο που να ταιριάζει σε όλους μας. Και το θέμα εδώ δεν είναι μόνο η τελικοί χρήστε είναι και θέμα ευαίσθητη τεχνολογίας. Θέλουμε να καταλήξει αυτή σε λάθος χέρια. Νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε από τις Ηνωμένε Πολιτείε στο θέμα αυτό, διότι όσον αφορά και τους τελικούς χρήστε και τις ευαίσθητες τεχνολογίες, ε, ε, εφαρμόζει πιο αυστηρού κανόνε από ότι εμείς. Επίσης, ε, δεν θα ήθελα να ονοματίσουμε συγκεκριμένες χώρες. μόνο σε μια περίπτωση, τις περιπτώσεις των χωρών που δεν πληρούν τις κοινέ προϋποθέσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε μια εξαίρεση. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες χώρες που δεν εφαρμόζουν τους κοινού κανόνες. Και ελπίζω ότι εδώ στις κοινέ μας συνεδριάσεις θα μπορέσουμε να βρούμε διατύπωση που να μπορούν να αποδεχτούν όλοι θα πρέπει να σκεφτούμε ότι εκπροσωπούμε τους πολίτες της, Ευρωπαϊκ... της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν εκπροσωπούμε τις κυβερνήσεις μας. Έχουμε μια συγκεκριμένη υποχρέωση ως κοινοβούλιο και σε αυτήν θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Πρόλαβα να συνομιλήσω με την ώρα από τους σκιώδεις εισηγητές. Δεν πρόλαβα να μιλήσω ακόμα με... Μπόρεσα να συνομιλήσω με κάποιους από τους ε, σκιώδεις εισηγητές, όχι όμως με όλους. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσω να το κάνω. Στις 22 Οκτωβρίου θα έχουμε συνάντηση σκιωδών εισηγητών. Στο μεταξύ θα λείπω δυστυχώς. Ε, σας ευχαριστώ όμως διότι με ενδιαφέρον διάβασα τις τροπολογίες σας και... Θα προσπαθήσουμε να βρούμε καλούς συμβιβασμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στους σκιώδεις εισηγητές. Ο κύριος Τουνέκελα είναι πρώτος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το βρίσκω πολύ θετικό που μπορούμε να μιλήσουμε έτσι με την εισηγήτρια και προσβλέπω στις συμβαστικές τροπολογίες τότε θα σκεφτούμε και θα αποφασίσουμε. Έχουμε χρόνο. Το ΕΛΚ πάντως ως κύρια γραμμή έχει ότι εκείνη η θέση πρέπει να έχει ένα θετικό αντίκτυπο. Να είναι δεσμευτική νομικά και συγχρόνως την τελική απόφαση να μπορούν να την πάρουν τα κράτη-μέλη. Αυτή η κοινή θέση είναι κάτι που εκτιμούν και τρίτες χώρες και έχουν συμφωνήσει. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να ελέγξουμε πολύ καλύτερα το παράνομο εμπόριο όπλων, το λαθρεμπόριο όπλων και να υπάρχει η ικανοποιητική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών μελών. Κυρίω αν κάποιες άδειε έχουν ακυρωθεί από μια χώρα μέλο, είναι πολύ σημαντικό οι άλλες χώρες μέλη να ενημερώνονται από αυτού. Αυτό που είναι επίση σημαντικό να έχουμε υπόψη μα είναι ότι τα όπλα δεν είναι κακά από μόνα τους. Εξαρτάται από τη χρήση. Εξαρτάται από το ε, τι θέλουν να πετύχουν αυτοί που τα κατέχουν και το κατά πόσο τηρούν τους κανόνες, τους νόμους ή όχι. Οπότε η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρίσκεται στην καρδιά της ευρωπαϊκής ε, κοινή πολιτικής ασφαλείας και άμυνας. Γι' αυτό λοιπόν ένας λόγος παραπάνω να, εφόσον την έχουμε, να αποφύγουμε την ε, μεγάλη εξάρτησή μας από αλλού όσον αφορά την αμήνυνά μας. Είναι σημαντικά τα όπλα γιατί δρούν αποτρεπτικά σε περίπτωση επίθεσης. Στην Ουκρανία, για παράδειγμα. Και συνεπώς αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να εξεταστούν κατά περίπτωση και σύμφωνα πάντα με την κοινή θέση. Όπως είπα, με ενθαρρύνει κοινή θέση της εισηγήτριας και προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία και καλή έκθεση τελικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κι εμείς. Η κυρία Ενέσα Γιάλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την κυρία Βαλέρο για το έργο της προσπαθεί στο διάλογο να συμπεριλάβει όλες τις ομάδες και προσπαθεί να προσεγγίσει τις θέσεις με συμβαστικές προτάσεις. Στην ομάδα μου όλοι είμαστε στη διάθεσή της. Θέλω να επιθυμίσω ότι για τη δικιά μου την ομάδα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι η έκθεση αυτή μιλάει για τον έλεγχο, έτσι, για τον έλεγχο των εξαγωγών το πλαίσιο της κοινή θέση λαμβάνεται υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια και σε περίοδους κρίσης έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά έχουν συμβεί πολλά. Οι εξαγωγές λοιπόν έχουν και άλλες πόρτες παράνομες και καλυμμένα. Οπότε πολλές φορές τα όπλα αυτά τα οποία εμείς εξάγουμε τελικά ξαναμπαίνουν από την πίσω πόρτα και παράνομα στην Ευρώπη. Δεν είναι ότι απλώς λέμε εξάγουμε όπλα, μένουνε δεν ξέρω εγώ πού μένουνε. Όχι, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη διπλή μας ευθύνη. Δηλαδή πρώτα απ' όλα σε ποιον εξάγουμε τα όπλα, με ποιες κυβερνήσεις δηλαδή έχουμε τέτοιο εμπόριο. Υπάρχουν αυτά τα κριτήρια στην κοινή θέση βέβαια, αλλά επιπλέον πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτές οι εξαγωγές πρέπει να έχουν διπλή κλίδα ασφαλείας για να μην επιστρέφουν παράνομα τα όπλα αυτά και ανεξέλεγκτα στις χώρες μας. Χαιρετίζουμε λοιπόν και χαιρόμαστε για την ε, προθυμία της εισηγήτριας να επιβεβαιώσει το θέμα της νομιμότητας στον έλεγχο και στις εξαγωγές τελικά των όπλων, ότι θα είναι πάντα στα πλαίσια της κοινή θέσης και βάση του δικαίου, της νόμιμης άμυνας δηλαδή. Και κατά τα άλλα για τα μη στρατιωτικά όπλα, ξέρουμε ότι για μερικές χώρες είναι κάτι σημαντικό λόγω νοοτροπίας. και ε, συνηθιών, όπως για παράδειγμα τα κυνηγητικά όπλα, που σε μερικές χώρες ε, κυκλοφορούν πολύ γιατί συνηθίζεται. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κρανσίντευσκη, θέλετε κάτι να, να προσθέσετε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απολύτως με αυτά που μόλις άκουσα και μπορώ κυρίως να συμφωνήσω με αυτό που άκουσα κυρίως από τον εκπρόσωπο του ΕΛΚ δηλαδή ότι μια κοινή θέση πρέπει να λάβει υπόψη την εθνική κυριαρχία. Οι εξαγωγές όπλων αφορούν αυτή ακριβώ την εθνική κυριαρχία. Είναι πολύ σημαντικό. Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να βρεθεί μία ισορροπία δίκαιη μεταξύ όλων αυτών των κοινών στοιχείων που θέλουμε να προσθέσουμε, από τη μία εξαγωγές όπλων και από την άλλη σεβασμό της συλλογικής άμυνας. Είναι δύο κύρια σημασία ε, στοιχεία και πρέπει να υπάρξει μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των δύο. Ένα ακόμη θέμα το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι αυτή η κοινή θέση πρέπει να εφαρμοστεί με ε, ομοιόμορφο τρόπο παντού. Από γεωγραφικής απόψεως εννοώ παντού. Και το λέω αυτό σε σχέση με, τα, με την κατάσταση τώρα στη Μέση Ανατολή εμείς στις τροπολογίες μας θα τονίσουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα κριτήρια αυτά που θέλουμε να ισχύσουν πρέπει να ισχύουν και για τους ε, ε, προσανατολάς ε, γειτονές μας και αναφέρομαι και στη Ρωσία. Δεν ισχύει πάντοτε αυτό. Η Ρωσία κατά καιρούς είχε ένα κατά τη διαφορετικό καθεστώς ε, και μιλάω τώρα για την κατάσταση με ε, τα Μιστράλ. Η Ρωσία είχε μία κάπως προνομιακή μεταχείριση και πρέπει να έχουμε κριτήρια τα οποία θα εφαρμόζονται με ισότιμο τρόπο, ομοιόμορφα, ώστε να μην υπάρχουν ε, προνομιακές μεταχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λόζινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν ήμουν παρούσα κατά την πρώτη συζήτηση. Η πολιτική μου ομάδα όμως και εγώ δεν έχουμε σημαντικές διαφωνίες σε σχέση με το σχέδιο της κυρίας Βαλέρο. Δεν ξέρω τι συμβιβασμοί θα προκύψουν από τις συζητήσεις, δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη για αυτό. αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι η κοινή θέση αποτελεί πολύ καλό πλαίσιο. Τα κριτήρια έχουν εκπονηθεί και κατά τη γνώμη μου το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστούν σωστά και αποτελεσματικά τα κριτήρια αυτά. Επικροτώ το σχέδιο έκθεσης ως έχει. Έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες. Στις 180 τροπολογίες εντύπωση μου έκανε ότι κάποιες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και ότι προσπαθεί να δοθεί διαφορετικό επίκεντρο στην έκθεση, κάτι που δεν θεωρούμε ότι ενδείκνυται. η, η συγγήτρια και άλλες δύο πολιτικές ομάδες από ό,τι γνωρίζω θεωρούν όπως και εγώ το άρθρο 10 της κοινή θέσης απαραίτητο. Και ελπίζω ότι οι τροπολογίες για το άρθρο 10 θα υιοθετηθούν στην ε, ε, έκθεσή σας. Αυτό ήταν σημαντικό θέμα για μας μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω σκιώδη εισηγητή του EFTD. Δεν είμαι σίγουρη αν ο κύριος Άφραζερ ήταν ε, ο σκιώδης εισηγητής της πολιτικής του ομάδας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, το ότι συμβαίνει κάτι μία φορά δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμβαίνει πάντοτε. Θα ήθελα ε, παρόλα αυτά να συμφωνήσω με τον συνάδελφο από το ΕΛΚ. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε την ελευθερία στα κράτη-μέλη Καταρχάς πρέπει να υπάρξει μία ε, κοινή απόφαση και αυτή η, η κοινή απόφαση πρέπει να είναι ανεξάρτητη της Ευρώπης συχνά. Οι κοινέ αποφάσεις μας ε, υπαγορεύονται από εξωτερικούς που δεν έχουν τίποτε να, δεν έχουν καμία σχέση με τα εσωτερικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλάω για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν, ε, είναι παράδεκτο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα δικά της συμφέροντα που δεν είναι ούτε του ΝΑΤΟ ούτε άλλων εξωτερικών φορέων. Δεύτερον, είναι πρέπει να είναι ε, απόλυτη η ελευθερία των κρατών μελών. Αυτή είναι η άποψή μα. Θεωρούμε σκανδαλώδη τον τρόπο με τον οποίο η Γαλλία ε, ενήργησε στην ε, υπόθεση Μιστράλ. Ε, είναι, είναι σημαντική ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία σε τεχνολογικό επίπεδο, και μιλάω για τη Γαλλία που είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης... που έχει μια τεχνολογική ανεξαρτησία, γιατί το είπα και για την Μεγάλη Βρετανία, η οποία δεν έχει τεχνολογική ανεξαρτησία εξαρτάται για ε, τα υποβρύχια της, ε, για, τα, για τις βόμβες της ε, απολύτως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς έχουμε όμως μια ανεξαρτησία και θέλουμε να τη διατηρήσουμε. Αυτή είναι η δική μας άποψη. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και για το μέλλον. Μιλάω για την τεχνολογική ανεξαρτησία. Επομένως, κοινή απόφαση ναι, υπό τον όρο βέβαια να υπάρχει μια πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά η ανησυχία που έχουμε εμείς ως ομάδα και για τη δική μας χώρα που εξακολουθεί να έχει μία ανεξαρτησία τεχνολογική να την διατηρήσει και να μην ε, ε, υποκύψει ε, στις επιθυμίες όλων γιατί η εθνική κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση προς την εισηγήτρια. Είπατε ότι η εφαρμογή της κοινή θέση δεν λειτουργήσε πάντα σωστά στην πράξη. Από ποιες πηγές έχετε λάβει αυτή την εκτίμηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο για τη σημερινή μας συνεδρίαση και καθότι δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των σκιωδών εισηγητών, προτείνω να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή για την έκθεση για τις εξαγωγές όπλων και την εφαρμογή της κοινή θέσης. Θα γίνει η συνάντηση των σκιωδών εισηγητών και θα εξετάσουμε τις τροπολογίες στις 12 Νοεμβρίου. Συμφωνούμε? Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. <coughs> Παρακαλώ κυρία Βαλέρο, έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τις παρεμβάσεις τους. Νομίζω ότι στις 22 Οκτωβρίου θα έχουμε μια παραγωγική συνεδρίαση και θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Γκάλερ ότι δεν ε, το λέει αυτό μόνο μία μελέτη. Έχουμε την έκθεση COARMS και θα πρέπει να την εξετάσουμε σε σχέση με τα όσα έχουμε κάνει στο παρελθόν. Είναι όμως ένα θέμα που έχω εξετάσει επί τρία χρόνια, τις εξαγωγές όπλων από τη Σουηδία και βλέπω σε τι βαθμό δεν έχουν γίνει αυτά που προβλέπει η κοινή θέση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα κλείσουμε το θέμα αυτό στην ημερησία διάταξη. Το επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη είναι η αντιμετώπιση του ακραίου εξτρεμισμού. Θα ήθελα να καλωσορίσω δύο ομιλητές. Το θέμα αυτό προτάθηκε από όλους τους συντονιστές, ιδιαίτερα όμως από τον κύριο Γκάλερ. Θα ήθελα λοιπόν να τον ευχαριστήσω για την πρότασή του και χάρη σε αυτήν ε, έχουμε εδώ τον κύριο Μαξούτ Κρούσε, εκτελεστικό διευθυντή του Διεθνούς Κέντρου Αριστείας για την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού, Χεντάια. Κατόπιν έχουμε την κυρία Χάνα Ντάνιελ, σύμβολο ε, στο πρόγραμμα καταπολέμησης του εξτρεμισμού. Όλοι ανησυχούμε λόγω του κύματος εξτρεμισμού που υπάρχει στις χώρες άμεσης γειτονίας. Είχαμε τα γεγονότα στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις σχετικά πρόσφατα. Είχαμε την τρομοκρατική επίθεση σε ε, χώρα υποψήφια για προσχώρηση, την Τουρκία. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να δώσω το λόγο στους ομιλητές μας. Κύριε Κρούσε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν από 40 χρόνια ένας ε, νέος Γερμανός έφυγε από το Βερολίνο και πήγε σε ένα μικρό μέρος στο Αμπιντάμπι που έγινε και η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Εμμυράτων μετά. Αγάπησε μία από τους Βεδοίνους και τελικά παντρεύτηκαν. Εγώ ήμουνα το νούμερο 2 των απογόνων τους. Όσοι γνωρίζουν την ιστορία μου, ρωτάνε πάντα το ίδιο. Μα λόγω τους ρωτάω, πώς θα με θεωρούσατε, Άραβα, Ευρωπαίο, άσπρο, μαύρο. Είμαι χριστιανός, είμαι μουσουλμάνος. Τι είμαι, ο Σοκράτης είχε πει ότι δεν είμαι Αθηναίος, δεν είμαι Έλληνας, είμαι πολίτης του κόσμου. Αυτό ακριβώς είναι η παγκοσμιοποίηση της ταυτότητας και αυτό ακριβώς είναι που απειλείται σήμερα. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι προωθούν το θάνατο, την καταστροφή. Εμείς όμως πρέπει να προωθήσουμε τη ζωή, την οτροπία της ζωής. Θέλουμε να χτίζουμε, όχι να καταστρέφουμε. Και αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε στο Χεντάγια, που είναι το Διεθνές Κέντριο Αριστείας για την Αντιμετώπιση του δύο Εξτρεμισμού, είναι ακριβώς αυτό. Θα σας εξηγήσω, είμαστε μια μικρή οργάνωση και θα σας αναφέρω κάποια στοιχεία κλειδί. Μετά ευχαρίστως να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχετε. Και η βοηθός μου, η Άιλα, θα με βοηθήσει με τις διαφάνειες. Το χεντάουα, λοιπόν, σημαίνει στα αραβικά καθοδήγηση. Έχει ισλαμική ρίζα. Δεν σημαίνει όμως γενικά καθοδήγηση. Το Σεπτέμβριο του 2011, όταν συνεδρίασε το Διεθνές Κέντρο για την του, της τρομοκρατίας, είχαμε πει ότι η ασφάλεια, η ανταλλαγή πληροφοριών για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας δεν φτάνουν. Ότι πρέπει να κοιτάξουμε βαθύτερα και την ψυχολογία και την κοινωνία, την οικονομία, την ιστορία και ακόμα και τη θρησκεία, είπαμε πιο πρόσφατα. Να δούμε ότι είναι περίπλοκο το φαινόμενο αυτό. Και αυτή ακριβώς ήταν η ιδέα από την οποία δημιουργήθηκε και το κέντρο μας, το ΧΕΤΕΧΑ και οι κόμικοι υπουργοί των ε, Ενωμένων Εμμυράτων αποφάσισαν ότι θα μπορούσε το κέντρο αυτό να έχει την έδρα του εκεί. Εκεί συμμετέχουν 29 κυβερνήσεις με ένα σύστημα περιτροπής ε, και ε, συνπροεδρίας. Δύο δηλαδή είναι πρόεδροι κάθε φορά. Βασιζόμαστε στην ιδέα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Χεντάια αποτελείται από τις 12 χώρες που συμμετέχουν στις διάφορες επιτροπές εργασίας. Είναι ένα μοναδικό μέρος γιατί εκεί κρατάμε ίσες αποστάσεις από όλες τις πολιτικές και από όλες τις ε, οργανώσεις αλλά και από όλα όσα κάνουμε. Με τη δομή μας έχουμε τρεις στόχους. Έρευνα και ανάλυση, αυτό είναι το ένα μας τμήμα. Έχουμε την κατάρτιση και έχουμε και τον διάλογο και τη συνεργασία. Το κάθε ένα από τα τμήματα αυτά βρίσκεται υπό την καθοδήγηση μιας διαφορετικής ε, κυβέρνησης. Ε, η Τουρκία στη μια περίπτωση, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι στην περίπτωση του διαλόγου και στο τρίτο τμήμα πρόκειται να έχουμε σύντομα ένα καινούριο επικεφαλής. Τι είναι αυτό το οποίο διαφοροποιεί το Χεντάγι, το κάνει μοναδικό. Πρώτον, είναι μια πολιτική οργάνωση χωρίς ιδεολογική τοποθέτηση. Δεν εξετάζουμε τα θέματα ιδεολογικά. Βασιζόμαστε σε γεγονότα, σε αποδείξεις. Δεύτερον, εμείς πιστεύουμε ότι όλοι είμαστε μέρος της λύσης. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε και με κυβερνήσεις αλλά και με κυβερνητικές ε, οργανώσεις γιατί όλοι συμμετέχουμε και όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε. Συγγνώμη αν σας βομβαρδίζω με την διαφοροποίηση. Τι είναι κάτι το πιο παραδοσιακό και κάτι είναι το πιο προθυμένο κέντρο αριστείας για την αντιμετώπιση των εξτρεμισμών. Εμείς πιστεύουμε ότι οι δάσκαλοι στα σχολεία αλλά και ειδικοί για την επικοινωνία, τα μέσα ενημέρωση, ή μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όλοι μπορούν να συνεισφέρουν για να βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα το φαινόμενο αυτό του βίου εξτρεμισμού. Εμείς έχουμε το εντοπίσει εννέα θέματα, δεν θα σας τα παρουσιάσω τώρα, τα βλέπετε εδώ, εξάλλου θα την έχετε την ε, παρουσίαση. Αλλά Τρία πράγματα θέλω να τονίσω. Πρώτον, ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης. Στην εκπαίδευση υπάρχει η λύση. Μερικές φορές βέβαια μπορεί να είναι και το πρόβλημα. Γι' αυτό και εμείς έχουμε εκπονήσει δύο έγγραφα. Το ένα είναι το Memorandum του Αμπουντάμπη με στοιχεία για την εκπαίδευση και τις καλύτερες πρακτικές σε αυτό το τομέα και θα υπάρξει και ένα ε, σχέδιο δράσης για τους συμμετέχοντες. Το δεύτερο θέμα που είναι πολύ σημαντικό και επίκαιρο είναι το θέμα των ξένων μαχητών. Λέμε δηλαδή πώς είναι δυνατόν κάποιος σε μια ξένη χώρα να ταυτίζεται με μια ξένη ιδεολογία και να πηγαίνει να ταξιδεύει τόσα χιλιόμετρα για να πάει να σκοτώσει κόσμο. Και τι κάνεις τότε, τι μέτρα, τι προληπτικά μέτρα για άλλα μπορεί να πάρει κανείς. Τέλος και με αυτό θα τελειώσω, είναι το θέμα της επικοινωνίας. Φυσικά και όλοι συμφωνούμε ότι οι ζωσπαστικές ομάδες σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρές. Δεν κάνουν απλώς προπαγάνδα, αλλά στρατολογούν τους νέους μας, τους παίρνουν από το φυσικό τους χώρο και τους πηγαίνουν σε έναν άγνωστο ξένο χώρο όπου τελικά καταλήγουν να σκοτώνονται. Με αυτά που σας λέω θέλω να καταδείξω με τι ακριβώ ασχολιόμαστε. Με αδερφές οργανώσεις στο Διεθνές Ινστιτούτο για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου δουλεύουμε προκειμένου να οικοδομήσουμε ε, δυνατότητες για να αντιμετωπιστούν αυτοί οι ξένοι μαχητές. Εμείς, επίσης, όλα αυτά έχουμε συζητήσει σε διάφορες συναντήσεις, συζητώντας ποιος κερδίζει από όλα αυτά και ποια μπορεί να είναι τα αποτελέσματα. 34 δραστηριότητες έχουμε συγχρόνως για αυτά τα θέματα με το Διεθνές Κέντρο Αριστείας για την Εντόπιση του Εξτρεμισμού και θέλουμε να δούμε πώς θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες προκλήσεις. Τέλος, θα ολοκληρώσω με το εξή. Σήμερα η Χεντάγια όσον αφορά την προβολή της δουλειάς μας και τη χρηματοδότηση που έχουμε, πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε χρηματοδότηση για διαφορετικά προγράμματα και ένα από αυτά χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσαμε έτσι να χρηματοδοτήσουμε 40 προγράμματα του χρόνου με 5 εκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση του δύο εξτρεμισμού. Ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές ε, τις εισαγωγικές παρατηρήσεις. Ε, δίνω το λόγο στην κυρία Χάνα Ντάνιελ. Ευχαριστώ. Καλημέρα και ευχαριστώ την Επιτροπή σας που με κάλεσε εδώ σήμερα να μιλήσω για το σημαντικό αυτό θέμα. Τονίζεται κάθε μέρα το θέμα του δύο εξτρεμισμού με ε, όλο και πιο αποτρόπες πράξεις κάθε μέρα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τις, ε, τους ε, βομβιστές αυτοκτονίες ε, στην Τουρκία και στο Ιράκ είχαμε άλλα περιστατικά και βλέπουμε ότι άλλος ένας Βρετανός πολίτης φεύγει από τη δημοκρατική μας κοινωνία για να προσχωρήσει στο Ισλαμικό κράτος. Όπως είπε ο προηγούμενος ομιλητής, ε, δεν ε, αρκεί να αντιμετωπίσουμε τη βία αποκλειστικά. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την ιδεολογία στην οποία βασίζεται. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ε, ιδεολογία μίσους που χρησιμοποιείται από το Ισλαμικό κράτος για να δικαιολογήσει τις ενέργειές της. Η ιδεολογία αυτή προωθεί την ιδέα του άλλου, ε, εμείς εναντίον των άλλων και ενθαρρύνει τον αποκλεισμό από την ευρύτερη κοινωνία. Και η μηχανή προπαγάνδας της ISIS προωθεί μετά ε, ε, μια θετική εναλλακτική λύση όπου οι μουσουλμάνοι υποτίθεται ότι μπορούν να ασκούν τη θρησκεία τους σε θηλυκό περιβάλλον. Και έτσι οι τρομοκρατικές ε, οργανώσεις ε, προχωρούν σε βίες πράξεις. Θα πρέπει λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό να εξετάσουμε το γιατί είναι τόσο αποτελεσματικό το μήνυμα της εξερμιστικής προπαγάνδας. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχουμε τις στρατιωτικές εικόνες ε, της, του ISIS και τις υποσχέσεις ενός ελεύθερου Ισλαμικού κράτους. Πολλοί θεωρούν ότι αυτές οι εικόνες είναι οι πιο βλαβερές, αλλά εξίσου βλαβερές μπορεί να είναι οι εικόνες υποστηρικτών του Ισλαμικού κράτους ε, που ζουν μια ειρηνική ζωή, τρώνε γλυκά, παίζουν στα πάρκα Αυτές οι εικόνες δείχνουν την ιδέα που θέλει να πουλήσει η ISIS, ότι θέλει να δημιουργήσει τέτοιες κοινωνίες. Και κανείς ε, δεν ε, αμφισβητεί τις ικανότητες ε, της ISIS στην προπαγάνδα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης. Και η Wall Street German λέει ότι η ISIS έχει παράγει φέτος 900 ε, μέσα προπαγάνδας, φυλάδια, εκπομπές κλπ. Και πολλά από αυτά έχουν να κάνουν ε, με το βιωτικό επίπεδο, με τη διατροφή, την, ε, το σχολείο και τέτοια. Το 50%, το 30% έχει να κάνει με στρατιωτικά θέματα και ελάχιστο κομμάτι έχει να κάνει με βίαιες πράξεις. Πώς λοιπόν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την προπαγάνδα που προωθεί την ιδεολογία και την βία. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις ελευθερίες ε, που έχουμε σε μια δημοκρατική κοινωνία και να τονίσουμε την ε, τρομοκρατική πλευρά του Ισλαμικού κράτους. Για παράδειγμα, τη μεταχείριση των γυναικών. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των θυμάτων ε, του Ισλαμικού κράτους είναι ε, μουσουλμάνοι. Ε, μεγάλο μέρος των μουσουλμάνων δεν συμφωνούν με τις δραστηριότητες, ε, δεν συμφωνούν με την ιδεολογία που δυσφημίζει τη θρησκεία τους και δημιουργούν αντι-ισλαμικά αισθήματα. Θα πρέπει να φροντίσουμε τα άτομα να έχουν τα μέσα που χρειάζονται για να επικρίνουν και να αντισταθούν στην προπαγάνδα. Και αυτό δεν είναι δουλειά μόνο των κυβερνήσεων. Θα πρέπει και μη κυβερνητικέ οργανώσει και ο ιδιωτικό τομέα να συμμετάσχουν στι προσπάθειε αυτέ. Εκστρατείε όπως η αλήθεια για την ISIS στο Twitter, ένα συνεχές ρεύμα που να δείχνει ε, ότι είναι ουτοπία αυτά που προβάλλει η ISIS, ε, είναι τρόποι να γίνει αυτό και οι πιο αποτελεσματικοί παράγοντες θα προέλθουν από την κοινωνία των πολιτών. Διότι είναι πιο αποτελεσματική η επιρροή των νομοτήμων. Και ενώ δεν θέλω να ε, το αναφέρω αυτό ως αποκλειστικά μουσουλμανικό πρόβλημα, ε, θα πρέπει να συνομιλήσουμε με τους ανθρώπους που βρίσκονται πιο κοντά στο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν ε, Υπάρχει επιφύλαξη μεταξύ ε, μετριοπαθών μουσουλμάνων να προβάλλουν μια εναλλακτική λύση. Θα πρέπει να φροντίσουμε οι μουσουλμάνοι να νιώθουν ε, ευπρόσδεκτοι. Ε, το Ισλάμ δεν είναι μόνο μια θρησκεία, είναι και μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, την οποία θα πρέπει να εκτιμούμε. Υπάρχει μια έκθεση που λέγεται 2000 και μία εφευρέσεις που δείχνει τον πλούτο του Ισλαμικού κόσμου από την Ισπανία μέχρι την Κίνα και 400.000 επισκέπτες είχε η, η έκθεση αυτή. Και ε, πρέπει να βοηθήσουμε οι μειονοτικές ομάδες να έχουν καλύτερη αντιπροσώπηση και να συμμετέχουν στα κοινά. Θα πρέπει να γνωρίζουν από πού προέρχονται και να ταιριάζουν στην κοινωνία στο σύνολό τους να ενσωματώνονται σωστά. Θα πρέπει επίσης να καταλάβουμε την ποικιλομορφία μεταξύ των ε, των μουσουλμάνων. Υπάρχουν 44, ε, εκατομμύρια μουσουλμάνοι στην Ευρώπη και δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι όλοι αυτοί ενίκουν στην ίδια κατηγορία. Ενώ κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι ο Ισλαμικός εξτρεμισμός είναι ένα ενιαίο κίνημα, ε, ουσιαστικά είναι πολλά διαφορετικά κινήματα. Και εμείς είμαστε μια δημοκρατική κοινωνία, αλλά υπάρχει μεγάλη επικοινομορφία ιδεών σε αυτήν. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό, ώστε να προωθήσουμε τα θετικά προγράμματα που υπάρχουν στις χώρες μας. Πρόσφατα, στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, έγινε η πρώτη διάσκεψη κορυφής κατά του βίαιου εξτρεμισμού και 75 ε, νέοι ακτιβιστές από διάφορες χώρες συμμετείχαν. Εγώ εντυπωσιάστηκα από τη δουλειά που προσπαθούν να κάνουν οι νέοι αυτοί άνθρωποι στις ε, κοινωνίες τους. Με ελάχιστους πόρους ε, και ελάχιστη κατάρτιση καταπολεμούν την εκτρεμιστική ιδεολογία και προβάλλουν εναλλακτικέ λύσεις. Τέτοιες πλατφόρμες στις οποίες συμμετέχουν νέοι από όλο τον κόσμο και όπου ενώνονται με κοινό στόχο την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού ε, είναι απαραίτητες για να φροντίσουμε ο εξτρεμισμός να μην συνεχίσει να απειλεί τις κοινωνίες μας. Επίσης θα πρέπει να ασχοληθούμε με τους τρόπους με τους ε, οποίους ε, προπαγανδίζει η ISIS. 90.000 tweets την ημέρα υπάρχουν συχνά από ε, την ISIS και η Europol κάνει πολύ καλή δουλειά, συνεργάζεται ε, με ε, τα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης όσον αφορά τις προϋποθέσεις χρήσης τους. Η ISIS έχει 46.000 λογαριασμούς Twitter και αποδεικνύει την αξία της τώρα η ιδέα ότι αν θέλουμε να προστατεύσουμε τους νέους από τον εξτρεμισμό θα πρέπει να επενδύσουμε αρκετούς πόρους στα κατάλληλα μέσα. Θα πρέπει να φροντίσουμε δηλαδή η εκστρατεία κατά του εξτρεμισμού να προβληθεί σωστά. Οι τρεις ιδέες που θα ήθελα να τονίσω εδώ είναι οι εξής. Καταρχάς, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το κίνητρο του βίαιου εξτρεμισμού είναι η εξτρεμιστική ιδεολογία. Αν ε, αφαιρέσουμε το κίνητρο, θα μπορέσουμε να αποφύγουμε και τον ε, βίαιο εξτρεμισμό. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, ένα θετικό αφήγημα το οποίο να αντίκειται ε, στην προπαγάνδα της ε, ISIS. Και επίσης ε, αυτό δεν είναι δουλειά αποκλειστικά για τις κυβερνήσεις, θα πρέπει να συμμετάσχει, να συμμετάσχει η κοινωνία των πολιτών και ο ιδιωτικός τομέας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ντάνιελ. Δίνω τώρα το λόγο. Ο κύριος Γκάλερ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις δύο ομιλίες σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για μας. και για τις χώρες από όπου έχουν ξεκινήσει αυτές οι προσπάθειες. Είναι μεγάλης σημασίας το ότι έχουμε οργανώσεις όπως η Χεντάια που εδρεύουν σε μουσουλμανικές χώρες. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στις δικές μας κοινωνίες. ώστε να ε, αποφύγουμε, να προλάβουμε οι πολίτες μας να πέφτουν σε τέτοιες ιδεολογικές παγίδες. Αλλά η ιδεολογία αυτή και τα διαπεριστατικά ανθούν συχνά σε Ισλαμικές χώρες. Θα πρέπει να εξετάσουμε τη διαφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης. Θα πρέπει να εξετάσουμε την σχέση ανάμεσα στο επίπεδο εκπαίδευσης και τα φαινόμενα αυτά. Ίσως ε, οι πλούσιες χώρες του αραβικού κόσμου να αποτελούν εξαίρεση, αλλά αν κοιτάξουμε την Τινησία και την Αίγυπτο, είμαι βέβαιος ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στο χαμηλό επίπεδο πολιτικού εξτρεμισμού και το επίπεδο εκπαίδευσης στην Τινησία. Νομίζω ότι στην Γεμένη είναι πολύ πιο ε, ευάλωτοι οι άνθρωποι απέναντι σε τέτοιες ιδεολογίες. Αυτό αποτελεί μια δική μου διαπίστωση. Γενικά, εντός των Ισλαμικών κοινωνιών θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος και αυτή είναι μια ερώτηση προς τις οργανώσεις σας. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Θα πρέπει να βρούμε θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ερμηνευτεί εκ νέου το Ισλάμ για τον 21ο αιώνα. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί δεν είμαστε μουσουλμάνοι. Θα πρέπει, δεν έχουμε την ε, ε, αξιοπιστία, δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Αλλά στα πανεπιστήμια, όπου εξετάζεται αυτή η θρησκεία, Πώς βλέπετε τις δυνατότητες να γίνει αυτό και πιστεύετε ότι οι εμπλεκόμενες κυβερνήσεις θα μπορέσουν να προωθήσουν κάτι τέτοιο ε, ή για παράδειγμα στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας να περιμένουμε ακριβώς το αντίθετο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σκάμ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα ευχα... επίσης να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω τους ε, δύο προσκεκλημένους μας σήμερα για τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα ε, η δουλειά του κέντρου Χεντάια. Είναι πάρα πολύ καλή πλατφόρμα αντιμετώπισης του βίαιου εξτρεμισμού. Αλλά θα ήθελα επί τη ευκαιρία να μάθω λίγο περισσότερα πράγματα. Θα κάνω μερικές ερωτήσεις συνεπώς, τις οποίες μπορείτε να ε, μας απαντήσετε για να καταλάβουμε περισσότερο. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μαθαίνουμε από τις καλές πρακτικές ε, γιατί είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα πλέον και συνεπώς πρέπει ε, σε παγκόσμιο επίπεδο να συνεργαστούμε. Βεβαίως υπάρχουν καλές πρακτικές και πρέπει να τις εντοπίσουμε και να τις ακολουθήσουμε. Προφανώς ε, υπάρχει αυτή η, μια Υπάρχει μια γραμμή που διαχωρίζει τον βίο με την ελευθερία ε, της ε, θρησκείας και πρέπει να δούμε πού ακριβώς θα την ε, τοποθετήσουμε αυτήν τη γραμμή. Ίσως λοιπόν θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο και το οικονομικό κομμάτι της όλης υπόθεσης. Προφανώς είναι γεγονός ότι από οικονομικής απόψεως σιγά σιγά γινόμαστε ένας κόμβος και πρέπει να ακολουθηθούν κάποια βήματα για να μπορέσουμε να, το, να παρακολουθήσουμε την κατάσταση. Το θέμα είναι αυτά τα βήματα, πόσο πολύ ε, έχουν αντίκτυπο στις άλλες χώρες και πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα βήματα αυτά ε, να μην ε, επηρεάζουν αθώους ανθρώπους και να μπλοκάρουν οι λογαριασμοί των ανθρώπων αυτών ακριβώς επειδή κάνουμε εμείς λάθος. Υπάρχει επίσης και το θέμα των πολιτικών ε, ζητημάτων που έχουν άμεση σχέση με αυτό το θέμα. Αυτοί οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν ε, το πρόσχημα της, ε, της θρησκείας και σε μερικές χώρες, όχι μόνο στην περιοχή αυτή αλλά και πέρα από την περιοχή, το χρησιμοποιούν ως εργαλείο για τους ε, δικούς τους πολιτικούς στόχους. Πώς κάνουμε τη διάκριση μεταξύ αυτών των δύο πραγμάτων, ώστε να μην συγχέονται τα πράγματα, αντιθέτως να μπορούμε να βοηθήσουμε. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σας πω, ακούσαμε όλο αυτό το θέμα των κοινωνικών μέσων δικτύωσης που μας είπε η Χάνα, τι εργασία και τι έρευνα έχετε ε, δει στο θέμα των μηνυμάτων, τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί ε, ο μανδύας ο θρησκευτικό που χρησιμοποιείται μέσω, υπάρχουν τα παραδοσιακά μέσα, υπάρχουν οι μάμιδες που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να περάσουμε κάποια μηνύματα. Και ένα ακόμη πράγμα που μας απασχολεί πάρα πολύ είναι το θέμα των ξένων μαχητών. Είναι σε μεγάλο βαθμό Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει εδώ. Τι είναι αυτό που τους κάνει από τη βολή αυτής της, ε, του μέρους που έχουν μεγαλώσει να πάνε σε μέρη όπου υπάρχουν τεράστια προβλήματα, βία και τεράστιες αντικσοότητες. Τι ακριβώς λοιπόν έχετε κάνει ως προς αυτό. Και Χάνα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω γιατί μας έφερες αυτήν την έκθεση ε, την οποία, στην οποία συμμετείχα και ε, την οποία δρομολόγησα εγώ στο Μάντσεστερ, μια πάρα πολύ ωραία πόλη. Είναι σημαντικό να τη φέρουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλη αυτή την ιδέα του πολιτισμού. Πολλοί μιλούν για τη σύγκρουση των πολιτισμών, ενώ στην πραγματικότητα είναι ότι όλοι οι πολιτισμοί συνδέονται συνδέονται μεταξύ τους και μάλιστα ο ένας ε, βασίζεται στον άλλον. Όλοι έχουμε συμμετάσχει σε αυτό. Το να έχουμε καλύτερη κατανόηση θα μπορέσουμε να, να, να μας βοηθήσει να, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και έχω ακούσει πάρα πολύ μεγάλη άγνοια και πολύ διαστρεβλωτικά πράγματα, ακόμη και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Συνοδάμσκι. Ο κύριος Κραντσινοντέμσκι. Έχω να κάνω μια ερώτηση προς την κυρία Ντάνιελ, γιατί, Ντάνιελ, γιατί Κάθε φορά που κάνουμε αυτή τη συζήτηση έχω την εντύπωση ότι κάτι λείπει, ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης ε, όσο υπάρχουν για παράδειγμα στις λογοτεχνίες, ε, στις συζητήσεις των ε, διανοωμένων για την, τις αιτίες και τις απαρχές της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης. Μήπως θα έπρεπε να κάνουμε και μεγαλύτερη αυτοκριτική γιατί γνωρίζουμε ότι ε, είναι πολύ πιο ελκυστικό πλέον αυτό το, το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης ε, Ίσως θα έπρεπε λοιπόν ε, να κάνουμε μία διάγνωση πιο βαθιά κοινωνική και να δούμε τι γίνεται στις κοινωνίες μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τι πάει λάθος και προκαλούν αυτήν τη ριζοσπαστικοποίηση. Όσο δεν το κάνουμε αυτό, πάντοτε θα υπάρχουν εκπλήξεις για μας. Ε, κάποιος, ε, για παράδειγμα, ε, στη Γερμανία, ένας πολίτης που έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Γερμανία, θα προσχωρήσει στο ISIS. Εγώ είδα στα, γερμανικά, στα γερμανικά πανεπιστήμια ε, πολλές γυναίκες διμένες με τον τρόπο που εκφράζει τη θρησκεία τους και δείχνει ενδεχομένως ότι υπάρχει μία τάση προς τον εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση. Δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε να έχουμε και μία πιο φιλοσοφική προσέγγιση. Ε, σχόλιο εκτό μικροφώνου από τον κύριο Τάνοκ δεν ακούμε δυστυχώ. Πάντω ο κύριο Κραζοντέμσκι συμφωνεί. Κύριε Τάνοκ, κοιτάξτε δεν ανοιχτή η συζήτηση λέει η πρόεδρο ε, κύριε Τάνοκ. Ε, δεν ε, ε, κάνουμε brainstorming. Μπορείτε να μας ζητήσετε το λόγο για να πάρετε το λόγο. Η κυρία Βαλέρο. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να είμαι σύντομη, διότι καλύφθηκα από τους προηγούμενους. Θα ήθελα να ρωτήσω, τι κάνετε για να έρθετε σε επαφή με το ευρύτερο κοινό. Αναφερθήκατε στα Εμμυράτα. Τι κάνετε εκεί και σε άλλες χώρες. Είδαμε ότι 5.000 ε, αλλοδαποί πολεμιστές ε, προέρχονται από την Ευρώπη, αλλά και από την Ινσία είδαμε χιλιάδες που πήγανε στην Συρία. Το μεγαλύτερο μέρος αλλοδαπών πολεμιστών λοιπόν ε, έρχονται από χώρες της Βόρειας Αφρικής. χρειάζεται ε, να προλάβουμε το πρόβλημα, αλλά πώς μπορούμε να μετρήσουμε την έκταση του προβλήματος ε, και, και το αποτέλεσμα των προληπτικών ε, ενεργειών μας. Όλοι θέλουμε να προλάβουμε, πώς θα το κάνουμε όμως και πώς θα έρθουμε σε επαφή με ε, τους σωστούς ανθρώπους, με αυτούς στους οποίους θέλουμε να απευθυνθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τονεκιέλα. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά πάρα πολύ ενθαρρυντικό αυτό το μήνυμα και πάρα πολύ ευπρόσδεκτο. Αναφέρατε σημασία τη σημασία της ταυτότητας και της εκπαίδευσης γιατί νομίζω η ταυτότητα και η κατανόηση της έννοιας και της σημασίας της ζωής είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικότερα για τους νέους ανθρώπους. Ε, δεν είναι περίεργο που πάρα, πολύ, ο, που πάρα μεγάλο το ποσοστό των νέων ανθρώπων που ενδιαφέρεται για αυτές τις εξτρεμιστικές λύσεις έχει να κάνει με το κατεστημένο, έχει με την κοινωνικο-οικονομική ε, ζωή ε, και κατάσταση να κάνει όλη υπόθεση και επίσης δεν καταλαβαίνουν τη σημασία της ζωής και έχει να κάνει νομίζω μερικές φορές και με τις πολιτιστικές τους ρίζες. Οπότε προσπαθούν με πιο σύντομο τρόπο να λύσουν τα προβλήματα της ζωής τους για να δει ε, ότι μπορούν να αντιταχθούν στο κατεστημένο. Ε, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά είπατε ότι η εκπαίδευση από μόνη της δεν αρκεί, ότι χρειάζεται μια καλύτερη, διεξοδικότερη εκπαίδευση και συμφωνώ αν Μιλάμε για κατανόηση μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών. Ε, δεν μπορεί να ε, αποφύγει κανείς τις βασικές αξίες ε, των θρησκειών. Ο κόσμος του Ισλάμ είναι πάρα πάρα πολύ στενά συνδεδεμένος με το θέμα της θρησκείας, ενώ ένα άλλο κομμάτι του κόσμου είναι περισσότερο γνωστικιστές. Οπότε κατά κάποιο τρόπο υπάρχει περίπτωση να προσβάλλουμε αυτό που είναι ιερό για τη θρησκεία. Και συμφωνώ απολύτως με το συνάδελφο που είπε ότι δεν είναι ξέχωρε οι θρησκείε. θα μπορούσαν να συμπληρώνουν και να εμπλουτίζουν η μία την άλλη. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο επί τη βάση αμοιβαίου σεβασμού. Αν μπορούσαμε να εμφυσίσουμε στο, στον συλλογισμό των ανθρώπων την ιερότητα και τη σημασία της ζωής, αυτό θα ήταν μία λύση. Ε, ελπίζω να μπορέσουμε να το κάνουμε, αλλά όπως είπα, το παράδειγμα σας είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Ευχαριστώ. Thank you, sir. Ευχαριστώ πολύ. Mm, thank you, Mr. Um, um, Cruz. Uh, Εσείς έρχεστε από μια διαμεσογειακή, ε, προσέξτε, προήλθατε από μια διαμεσογειακή σχέση, εγώ από μια διατηρητική σχέση. Ε, νομίζω ότι έχουμε μια προνομιούχο θέση και έχουμε ένα καθήκον να κάνουμε κάτι βάσει της ιδιότητάς μας αυτής. Δεν είναι όλος ο κόσμος ευχαριστημένος προφανώς. Αν γίνομαι πάρα πολύ Αμερικανός, ο κύριος Αφουσέρ δεν θα χαρεί καθόλου. Αν γίνω πάρα πολύ Ισπανός... Ε, κάποιος ε, επίσης μπορεί να δυσαρεστηθεί. Οπότε έχουμε τέλος πάντων αυτό το ιδιαίτερο προνόμιο επειδή ακριβώς ε, ε, είμαστε ένα μείγμα, πρέπει να προσπαθήσουμε να συμφιλιώσουμε και δύο διαφορετικούς πολιτισμούς. Γνωρίζω μερικά πράγματα για τη δουλειά σας και με ενδιαφέρει για τη χώρα σας και νομίζω ότι ο συνάδελφος ε, το είπε ήδη ε, ότι είναι πολύ σωστά τα βήματα που γίνονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το θέμα είναι όμως ότι ε, είμαστε στο μέτωπο μιας πάρα πολύ μεγάλης μάχης και δύσκολης μάχης ενάντια στον εξτρεμισμό και εσείς είστε στην πρώτη γραμμή της μάχης αυτής. Συγχαρητήρια λοιπόν για τη χώρα σας και στην περίπτωσή σας κιόλα με το ε, ίδρυμα αυτό, το Ινστιτούτο αυτό, θα ήθελα να σας πω ορισμένα ε, πράγματα, να σας ρωτήσω ορισμένα πράγματα για να εμβαθύνετε παραπάνω. Το ερώτημα Τη εκπαίδευση ε, που το έθεσε και ο συνάδελφο και πράγματι δουλεύετε κι εσεί πάνω σε αυτό. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε τις αιτίε, τις ρίζες του προβλήματος και κάτι το οποίο επίση συμβαίνει στην Ευρώπη και, θα ήταν χρήσιμο να τα ακούσουμε είναι η απορρίζωστη παστικοποίηση ε, στις φυλακές που μερικές φορές ε, συμβαίνει και αυτό. Μπορεί να πηγαίνει κάποιος, ε, μπορεί να πηγαίνει κάποιος στη φυλακή και τελικά να καταλήγει εξτρεμιστής γιατί εκεί κάνει αυτή την αλλαγή προς τον εξ, εξτρεμισμό. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα, μια ρητορική ερώτηση. οι διπλές ταυτότητες. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Και εγώ θα ήθελα να δώσω μια έτσι απλή απάντηση. Αν είσαστε από μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήκος δηλαδή, έχετε αυτή την υπηκότητα και είσαστε και Ευρωπαίος. Αν είσαστε κάποιος μουσουλμανικής προέλευσης, αλλά εδώ και δύο-τρεις γενιές ζείτε στην Ευρώπη, έχετε αυτό το πρόβλημα, δηλαδή να είσαστε ανάμεσα σε δύο με το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί. Όσον αφορά την υπηκότητα, βέβαια είναι ξεκάθαρο. Τα υπόλοιπα είναι πιο πολύ κοινωνιολογικά. Και έτσι έρχομαι και στο δεύτερο, στο θέμα της εκπαίδευσης. Θα σας δώσω ένα γερμανικό παράδειγμα. Στη Γερμανία, προς το παρό, δεν είχαμε Ισλαμικό, Ισλαμική τρομοκρατία. Οι περισσότεροι μετανάστες που είναι στη χώρα μου προέρχονται από την Τουρκία, που είναι ένα κοσμικό κράτος, μη θρησκευτικό προσπαθούμε κι εμείς να εκπαιδεύσουμε τους ημάμιδες, τους Τούρκους στη Γερμανία και για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτοί οι μουσουλμάνοι οι ημάμιδες στη Γερμανία να ε, παραμείνουν σε αυτό το κοσμικό πλαίσιο. Όχι ότι δεν θα μπορούσαν να ασκούν τη θρησκεία τους, αλλά να μην ξεχνάνε ότι είναι στα πλαίσια ενός κοσμικού κράτους. Η Τουρκία λοιπόν, ναι, μεν ε, έχει ως θρησκεία τη μουσουλμανική θρησκεία, αλλά είναι ένα κοσμικό κράτος. Αυτό είναι και το δικό μας μοντέλο στην Ευρώπη στο κάτω-κάτω. Έχουμε το χριστιανισμό ως θρησκεία, αλλά είμαστε κοσμικά κράτη. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή αυτή η διάκριση ανάμεσα στη θρησκεία και το κράτος. Και το μήνυμα το μουσουλμανικό που εκπέμπεται θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, να ξεκαθαρίζεται. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσω της εκπαίδευσης. Αυτή η διάκριση και αυτή η σχέση ανάμεσα στα δύο, το κράτος και τη θρησκεία. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κρούζετ να απαντήσει και να πει τις δικές του απόψεις. Ο κύριος Κρούζετ λοιπόν πρώτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρεις σελίδες έχω γράψει εδώ με τις υπέροχες ερωτήσεις και σχόλιά σας. Θα προσπαθήσω λοιπόν να τα συγκεντρώσω και συγγνώμη εκ των προτέρων να ξεχάσω κάτι. Εννοείται η επικοινωνία παραμένει. Αρχίζω πρώτα με το δικό σας ερώτημα τι γίνεται από τη μουσουλμανική κοινότητα στον Ισλαμικό κόσμο, τι πρέπει να κάνει ακόμα. Εγώ φυσικά δεν μπορώ να απαντήσω εκ μέρους της ε, αλλοχωρών και οργανώσεων. Το βέβαιο είναι, και θα σας δώσω τα εξή παραδείγματα. Πρώτον, υπήρξε μια πρωτοβουλία για να δημιουργήσουμε κάτι που είναι η πρόθεση της ειρήνης με μουσουλμανικά φόρουμ. Ε, δουλεύει εδώ και δύο χρόνια ειναι ενα ένας Ισλαμο-Ισλαμικός διάλογος, εσωτερικός δηλαδή μέσα στο Ισλάμ, κατά του ριζοσπαστικού Ισλάμ. Είναι μια εσωτερική διαδικασία λοιπόν που υπάρχει στον Ισλαμικό κόσμο και εμείς είχαμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε ένα βαθμό. Δεύτερη πρωτοβουλία είναι το Μουσουλμανικό Συμβούλιο. Εδώ ηγούνται διάφορες ηγετικές προσωπικότητες, ε, μάμιδες και άλλοι του μουσουλμανικού κόσμου. Η ιδέα είναι να επιτρέψει την ανταλλαγή απόψεων σε θεολογικό επίπεδο ώστε να ενισχυθεί η σύγχρονη Ισλαμική σκέψη σε αντιπαράθεση με την πιο παραδοσιακή. Πρόσφατα τα Εμμυράτα και άλλοι στα πλαίσια της συνεργασίας ε, της Διεθνούς κατά της ΔΑΣ έκανε το κέντρο Πασαγουάπ. Τι είναι αυτό? Είναι μία online πρωτοβουλία προκειμένου να αποδομεί κάθε φανατικό μήνυμα και να φέρνει στην επιφάνεια στην πράξη τι γίνεται. Είναι μηνύματα και χαιρόμαστε πολύ που και εμείς συμμετείχαμε στην δημιουργία του. Επικεντρώνεται στην εξή απλή ιδέα. Το πρόβλημα, και έτσι έρχομαι στη δεύτερη ερώτηση που έχει να κάνει με την έκφραση και τα κοινωνικά δίκτυα, την ελευθερία έκφρασης κλπ. Και πώς θα καταπολεμήσουμε έτσι τον εξτρεμισμό. Θέλω να είμαι ειλικρινή. Σε διάφορες συναντήσεις που πήγα, κάποιοι κυβερνητικοί παίρναν το κινητό, το σηκώνανε, το δείχνανε σε όλους και λέγανε αυτό δεν είναι κινητό, αυτό είναι ένα όπλο. Γιατί με τα κινητά γίνονται επιθέσεις στις κοινωνίες. Ωραία, και εγώ μπορώ να πω να αυτό είναι ένα μολύβι, αν το βάλω στο μάτι κάποιου, βεβαίω και θα είναι κακό. Τώρα είναι κακό όμως το μολύβι από μόνο του. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι όταν η μικρή μου αδερφή και τα αδέρφια μου 6, 7, 15 τη νύχτα ξυπνούν και πάνε στην ε, αυτοριζοστικοποίηση, κανένας δεν τους στρατολογεί. Συνδέονται. Πώς συνδέονται όμως και τι είναι αυτό που τους κάνει να περάσουν στο επόμενο βήμα. Αυτό το δεύτερο βήμα είναι αυτό που θέλουμε, πάνω στο οποίο θέλουμε να δουλέψουμε. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Είναι η πραγματικότητα. Έχουμε κάποιο κενό. Κάποιες ομάδες έρχονται με κάποιες υπέροχες φωτογραφίες παιδιών. Έρχονται με φωτογραφίες θυμάτων και μας λένε δεν κάνατε τίποτα. Θέλετε να κάνετε τη διαφορά, Έχει, θέλετε κάποιο σκοπό, ελάτε μαζί μας και θα το πετύχετε. Αυτό λένε. Πρέπει εμείς λοιπόν να αποκτήσουμε τη δυνατότητα να αντισταθούμε σε αυτό, να έχουμε έναν άλλο λόγο για να το παρακάμψουμε. Έρχομαι και στις άλλες σημαντικές σας ερωτήσεις. Η συζήτηση για την θρησκεία από τη μια και την πολιτική δράση από την άλλη. Όλοι το γνωρίζουμε και είναι πρωταθλήτρια η Ευρώπη, ότι είναι μια συζήτηση που συνεχίζεται. Υπάρχουν ομάδες που πάντα λένε η δική μου η πίστη έχει κάτι να πει για τα δημόσια ζητήματα και θέλω να το κάνω. Ο Ζων Σακορισό, ο Βολτέρ και τα λοιπά. Προφανώς τώρα ε, γυρίζω στους τάφους τους με τέτοιες ιδέες. Αλλά υπάρχουν και στην Ευρώπη αυτές οι ιδέες και στη δημοκρατία. Και εντάξει, η συζήτηση καλά κάνει και συνεχίζεται. Και γι' αυτό και λέω ότι ήταν πολύ ωραίες οι ερωτήσεις σας. Αυτό το οποίο λείπει σήμερα είναι ότι δεν μπορούμε να γεννήσουμε νέες ιδέες που είναι αναγκαίες στους σύγχρονους καιρούς που ζούμε. Δεν είμαστε στην περίοδο τη σύγκρουση των πολιτισμών. Όχι, χτίζουμε πολιτισμό, συνδέουμε πολιτισμούς και περνάμε στο επόμενο στάδιο. Όταν λοιπόν κάποιοι μου λένε, ξέρεις εσύ είσαι μουράτη. Ε, όχι, εγώ είμαι κατά το ίμιση Γερμανός, είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει. Ότι είσαι από τα Εμμυράτα δηλαδή. Και άλλοι που μου λένε, μα εσύ είσαι Γερμανός, λέω όχι, είμαι κατά το ίμιση από τα Εμμυράτα. Σήμερα είπα σε κάποιον ακριβώς και γι' αυτό μπορείς να πεις ότι είμαι μισή καμήλα και τίποτα, τι θες να κάνω δηλαδή. Η... Αντίθετα με εσάς, κύριε Λόπες, μπορεί να μην μοιάζω με εσάς, αλλά έχουμε αυτό σεβασμό και βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Θέλω να κάνω και δύο σχόλια και ζητώ συγγνώμη γιατί πολύ θα ήθελα να συζητήσουμε περισσότερο για αυτά. Είναι το εξή. Πρώτο, η κριτική ανάλυση της συνεχιζόμενης συζήτησης στην Ευρώπη και στις μουσουλμανικές ε, κοινωνίες. Είδαμε τι έγινε με το Σαρλί Επτό. Συγκλονιστήκαμε όλοι. Γιατί ο υπεύθυνο ήταν κάποιος ο οποίος βρισκόταν σε ένα χώρο ο οποίος ήταν ε, το αποκορύφωμα της ελευθερίας. Κι όμως ήταν τόσο απελπισμένος να εκδηλώσει τη διαφωνία του που πήγε και σκότωσε κάποιον. Δηλαδή δεν ερχόταν από μια ύποπτη χώρα, από μια κατασταμένη χώρα, δεν ξέρω τι. Όχι, τη Γαλλία. Γιατί, τι λείπει λοιπόν εκεί. Τι δεν έχουμε δει καλά. Δεύτερος λόγος που συγκλονιστήκαμε. Τα θύματα, ένας από αυτούς ήταν από την ίδια κοινότητα. Ένα αστυνομικός που ήταν εκεί επίσης προερχόταν όπως και ο δράστης και ο οποίος αυτός ο θύλακας προστάτευε αυτόν που παραδοσιακά εντό αγωγικών είναι εχθρός. Το ερώτημα παραμένει. Όλοι αυτοί μεγάλωσαν στον ίδιο χώρο. Έδρασαν όμως διαφορετικά. Ο ένας σκοτώνει, ο άλλος προστατεύει. Και ο τρίτος λόγος που συγκλονιστήκαμε ήταν, και εδώ θέλω να είμαι ειλικρινής και με τον εαυτό μου και με όλους σας, το πραγματικό ζήτημα είναι το εξή. Τα συστήματά μας σήμερα. Μήπως έχουν αποτύχει να μας οδηγούν στην ταυτότητα αυτή που θέλουμε. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να μην βλέπουμε το χρώμα, να βλέπουμε τα υπόλοιπα, από όποιο και αν προέρχεσαι, ό,τι προσανατολισμό και αν έχεις, ό,τι πολιτικές απόψεις και αν έχεις. Το πραγματικό ζήτημα είναι αυτό, ανεξάρτητα από τις απόψεις, από τη φιλοσοφία σου, από το παρελθόν σου, τη θλίψη σου κτλ πώς μπορείς να δικαιολογήσεις την χρήση βίας απέναντι σε αθώος. Δεν έχει σημασία από πού ερχόμαστε. Όλοι είμαστε διαφορετικοί. Και εγώ ο ίδιος. Και ίσως γι' αυτό και ασχολήθηκα με την ψυχολογία. Και χαίρομαι που υπάρχουν και άλλοι ψυχολόγοι εδώ στην αίθουσα. Για μας είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Αλλά είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα. Και όπως είδατε και από την παρουσίασή μου έχουμε εννέα θέματα και θα έχουμε και περισσότερα στο μέλλον. Το τελευταίο, στο οποίο θέλω να αναφερθώ και θα ολοκληρώσω με αυτό, είναι το θέμα της εκπαίδευσης. Ειλικρινά μου αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις, γιατί αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι το εξή. Μπορώ να πω ότι η ΝΤΑΣ, η Αλκαΐντα είναι εγκληματικές οργανώσεις, η ΦΑΡΚ στην ε, Κολομβία, ΕΤΑ στην Ισπανία. Το θέμα είναι όμως ότι βάζω τίτλους και δεν δίνω τα μέσα, τα εργαλεία για επικριτική σκέψη. Ξεχνάω ότι η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι μόνο η γνώση, είναι και η κοινωνική σχέση, η σχέση με τις οικογένειές μας και οι κανόνες. Η εκπαίδευση λοιπόν είναι μια εμπειρική διαδικασία. Δεν είναι ότι ένας μιλάει και άλλος ακούει. Αυτός που ακούει και αυτός από τη δικιά του μεριά συμμετέχει σε μια διαδικασία επικριτικής σκέψης που θα το βοηθήσει να οριμάσει. Ευχαριστώ πολύ και ό,τι ερωτήσει άλλε υπάρχουν, είμαι στη διάθεσή σα. Πρόεδρο, λυπούμε, αλλά θα είμαι δύσκολη εδώ. Γιατί βλέπετε, έχουμε και το επόμενο πάνελ. Η κυρία Ντάνιελ όμω να απαντήσει και εκείνη παρακαλώ σε ερωτήσει και τα σχόλιά τη θέλουμε. Θα είμαι σύντομη. Θέλω κι εγώ να απαντήσω σε ερωτήσεις και συγγνώμη αν κάτι ξεχάσω. Ένα από τα πρώτα που ρωτήσατε είναι η σχέση της ζωσπαστικοποίησης με το επίπεδο ζωής. Νομίζω ότι απλοποιούμε πάρα πολύ το θέμα αν πούμε ότι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο με ζωσπαστικοποίηση είναι αυτοί που έρχονται από πιο χαμηλά επίπεδα διαβίωσης. Όχι. Πριν από λίγους μήνες, τρία κορίτσια πήγαν από το Ανατολικό Λονδίνο στη Συρία δεν προέρχονταν από φτωχές οικογένειες, ήταν φοιτήτρε. η μία θα πήγαινε και στο Οξφόρδη. Άρα είχαν επιλογές, δεν είναι ότι δεν είχαν και όμως αποφάσισαν να πάνε στη Συρία. Όσον αφορά το μήνυμα και την ερμηνεία του τον 21ο αιώνα. Εγώ δεν είμαι σε θέση και δεν νομίζω ότι είναι κανείς. Πάντως, δεν νομίζω ότι πρέπει να ξαναγίνει. Από ό,τι βλέπω υπάρχουν μετριοπαθείς ε, μουσουλμάνοι και ομάδες που το κήρυγμά τους είναι μετριοπαθές. Πρέπει να τους βοηθήσουμε λοιπόν και να τους δώσουμε το κατάλληλο φόρουμ για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με θετικό τρόπο την ε, τρομοκρατία. Τον αγώνα μάλλον κατά της τρομοκρατίας βέβαια. Πώς φτάνουμε στον κόσμο χρειαζόμαστε τις κατάλληλες δομές. Γίνονται πολλά με τους μετροπαθείς μουσουλμάνους. Μπορεί να μην τα διαβάζουμε στην εφημερίδα κάθε μέρα, κάνουν δουλειά όμως και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει να εντοπίσουμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι ομάδες και να τις βοηθήσουμε. Δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε όμως, δεν πρέπει να τους λέμε εμείς τι να κάνουν, αλλά να διασφαλίσουμε ότι έχουν τους πόρους, τη στήριξη που χρειάζονται για να κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Για το θέμα της εκπαίδευσης, συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να κάνουμε πολλά και με τους ε, κοινωνιολόγους και κοινωνικές λειτουργούς. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να συζητιώνται στις τάξεις, στις κοινότητες και να υπάρχουν τα εργαλεία με καλές ε, μεθόδους και με προσοχή να μην ε, προσβάλλεται κανείς. Κάποιοι νέοι πράγματι ψάχνουν για νόημα στη ζωή τους. Αυτό όμως που θέλουν να ξέρουν είναι ποιος είναι ο ρόλος τους στις κοινωνίες που ζουν. Θέλουν να ξέρουν πώς μπορούν να συνεισφέρουν. Και εδώ είναι που μπορούμε να του στείλουμε ένα θετικό μήνυμα. Να μην είμαστε αρνητικοί. Μπορούμε να τους πούμε ότι σε νέος έχεις αξία, σε θέλουμε. Αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο προσκεκλημένους ομιλητές μας, τον κύριο Κρούζο και την κυρία Ντάνιελ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή. Πιστεύω και πιστεύω ότι μιλώ εκ μέρου όλων των συναδέλφων τη Υποεπιτροπή Άμυνα και Ασφάλεια ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό και βεβαίω θα λάβουμε υπόψη και αυτά που μα είπατε. Σα ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σα εδώ σήμερα. Θα παραμείνουμε σε επαφή και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επί του θέματος αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε ευθύ αμέσως στο επόμενο σημείο της της διάταξης. Επιτρέψτε μου απλώς να αποχαιρετήσω τους προσκεκλημένους μας. Ladies and gentlemen, please be... Κυρίες και κύριοι παρακαλώ καθίστε. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, παρακαλούμε να το κάνουν ήσυχα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι χαρά μου να καλωσορίσω τον στρατηγό Πατρίκ Τερουζιέ, ο οποίος μας είναι γνωστός, είναι ο πρόεδρος της Στρατιωτικής ε, Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης και το θέμα της συζήτησής μας, ε, επειδή πρόκειται για ανταλλαγή απόψεων με το στρατηγό, είναι η πρόοδος ε, της κοινή πολιτικής ε, άμυνας και ασφάλειας ε, τα τελευταία τρία χρόνια. Δυστυχώ, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, δεν θα ήθελα να χρονοτριβήσω περαιτέρω και θα ήθελα ε, στρατηγέ να σας δώσω ευθύς αμέσω το λόγο για να μας κάνετε τα εισαγωγικά σας σχόλια. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Ε, κάνετε μια δουλειά που είναι πάρα πολύ σημαντική στην Επιτροπή σας ε, και είναι πάντοτε πάρα πολύ εμπλουτιστικέ οι συζητήσεις με πάντοτε με πολύ χαρά έκανα συζητήσει μαζί σας. Ε, ξέρω ότι πριν από ένα μήνα ο Γενικός Διευθυντής του Γενικού Επιτελείου ήταν μαζί σας και συζητήσατε μαζί του το Κέντρο Επιχειρήσεων της Αταλάντας ε, στις 6 Νοεμβρίου αναλαμβάνει ο, έχω αναλάβει εδώ και τρία χρόνια ε, τον ρόλο του Προέδρου της Στρατηγικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, που συγκεντρώνει τους αρχηγούς ΓΕΔΑ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα να σας κάνω ένα μικρό απολογισμό, να αρχίσω καταρχάς από τις επιχειρήσεις, γιατί είναι το επίκεντρο της δουλειάς μας, αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω δύο ακόμη τομείς πολύ σημαντικούς. Ο πρώτος είναι η ανάπτυξη υποδομών, η προετοιμασία της συνεργασίας, του εξοπλισμού, των ε, δυνατοτήτων που έχουμε να εμπλακούμε συλλογικά ε, είτε σε επίπεδο 28 είτε σε πιο περιορισμένες συνθέσεις για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη των υποδομών ε, γιατί ε, συνεργαζόμαστε με, στενά με την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, Άμυνα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τον Ριορέντο Μεκ και την προκάτοχο συνάδελφό του, με τους οποίους ήμουν σε επαφή εχθές και με τους οποίους έχω τακτικές επαφές. Έχουμε βέβαια και κάποιους περιορισμούς ε, διότι μας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια ανάπτυξη υποδομών σε κάθε κράτος μέλος. Υπάρχει το θέμα του στρατηγικού διαλόγου επίσης. Εντός τριών ετών ε, είχα πολλές φορές διάλογο ε, στρατηγικής φύσεως κατόπιν ετήματος της ΥΠΑ της εκπροσώπου σε πάνω από 25 χώρες σε όλες τις επίρους και αυτό γιατί ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολιτική δομή και πολιτικός φορέας είναι γνωστή και αναγνωστή και εισακούεται και όλο και περισσότερο ε, και αυτό έχει έχει ως αποτέλεσμα να συζητώ με την Αφρική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, με την Κίνα, ε, όπου έκανα τον πρώτο στρατηγικό διάλογο με τον ομόλογο μου τον Κινέζο, όπως επίσης με την Ιαπωνία, με τη Νέα Ζηλανδία και με το σύνολο των φορέων ε, που δραστηριοποιούνται στον Ινδικό ωκεανό. Επομένως, ε, ο στρατηγικός διάλογος είναι πάρα πολύ σημαντικός και πολύ δυναμικός κατά τα τελευταία τρία χρόνια. Φτάνω τώρα στους ε, τις επιχειρήσεις. 230.000 στρατιώτες ε, σε ε, ε, πολλές επιχειρήσεις. Αυτό βέβαια σέβεται την, διαφορετική συμμετοχή από κάθε κράτος μέλος. 60 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια ευρώ τα οποία διαχειριζόμαστε βάσει της κατανομής αυτής ανάλογα με το κράτος μέλος. Είναι αποτελεσματική, είναι αφοσιωμένοι, αντιμετωπίζουν την πειρατεία, η σταθεροποίηση των χωρών που όπου υπάρχουν ε, πιέσεις, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Βαλκάνια, υποστήριξη ε, καθοδήγηση ε, των περιοχών όπου αντιμετωπίζονται τρομοκρατικά, τρομοκρατικές απειλές ε, ή υπάρχουν πολεμικές συγκρούσεις στη Σομαλία, στην οποία είχα πάει πριν από 10 ημέρες και σε άλλα μέρη της Αφρικής αντιμετώπιση και καταπολέμηση των, των δικτύων των εγκληματικών που δημιουργούν προβλήματα στα θαλάσσια ύδατα με την επιχείρηση Σοφία που θα τη γνωρίζετε πολύ καλά. Είναι πολύ καλή η διοίκηση των επιχειρήσεών μας. Θέλουμε επιτόπου να υπάρχει αποτέλεσμα βέβαια ε, έχοντας υπόψη τους περιορισμούς που έχουμε και να υπάρχει μια δυναμική πολύ θετική. Όμως ε, υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις ακόμη. Στην ε, κεντρική Αφρική νομίζω ότι μια μεγάλη πρόκληση είναι να καταφέρουμε να προκαλέσουμε τη μεταρρύθμιση, τη μετάβαση αυτό ε, με έχοντας υπόψη βέβαια το κέντρο των ε, δυνάμεων της ε, κεντροαφρικανικής δημοκρατίας που πρόσφατα έδειξαν ότι δεν έχουν καταλάβει ότι ε, οι στρατικές δυνάμεις πρέπει να εξυπηρετούν σε κάποιο βαθμό την πολιτική κατάσταση και είναι κάτι το οποίο οδήγησε στην επιχείρηση που έχει αρχίσει εκεί. Πρόκειται λοιπόν για μια πρόκληση η οποία σημαίνει κατά τη γνώμη μου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή. Τώρα, το πρόβλημα είναι τι θα κάνουμε μετά το 2016. Φτάνουμε στο τέλος ε, της ε, ε, επιχείρησης το θέμα είναι τι θα κάνουμε μετά. τι θα κάνουμε μετά, αυτό είναι το θέμα. κάνουμε πάρα πολύ σημαντική δουλειά για μένα είναι ένα, μία από τις μεγάλες επιτυχίες ε, και η άλλη επιτυχία είναι η επιχείρηση στον Ειδικό Ωκεανό. Στη Σομαλία ε, κάθε έξι μήνες, ε, ίσως και τέσσερις, ε, γίνεται αναθεώρηση για να ε, δούμε πώς έχει υπάρξει, αν έχει υπάρξει πρόοδος και από απόψεως ασφάλειας, αλλά και από απόψεως παρουσίας διεθνών φορέων. Βλέπω, ας πούμε, ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες πρεσβείες στη Μογκαντήσου σε σχέση με πριν από τρία χρόνια. Υπάρχει επίσης χρηματοδότηση από την Τουρκία, από άλλες χώρες του Περσικού κόλπου, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, εξαιρετικά υγιές γιατί δίνει τη δυνατότητα στην οικονομική ζωή να αναβιώσει. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπουμε σιγά σιγά ε, στη Σομαλία ότι αρχίζει να υπάρχει μια κάποια ηρεμία, όμως έχει ακόμη πάρα πολύ δρόμο, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι ε, να μπορέσει να ηγηθεί της επιχείρηση της Αμισόμ που είναι η μόνη που ε, εξασφαλίζει την ασφάλεια στην περιοχή. Και για μας αυτό είναι το θέμα ε, το οποίο θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι υπουργοί μας. Τι ακριβώς θα κάνουμε ε, πέρα από το Μογκαντήσου, τι στήριξη θα ε, παρέχουμε σε πλαίσιο στρατιωτικό, η Αλτέα, η επιχείρηση αυτή, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, είναι μία από τις επιχειρήσεις μας. Γνωρίζετε ότι ένα έγγραφο εταιρική σχέσης, ε, μια επίσημη εταιρική σχέση συνυπεγράφει μεταξύ της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα πρέπει να τη συνοδεύσουμε προοδευτικά ώστε να μπορέσει να συμμετέχει και αυτή στις επιχειρήσεις μας. Υπάρχουν και φήμες ότι η Βοσνία Ζεγοβίνη μπορεί να είναι υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι μια πρόκληση πώς είναι δυνατόν να διατηρήσουμε μια εκτελεστική επιχείρηση στην περιοχή με μια χώρα που είναι υποψήφια για ένταξη στην Ένωση. Αλλά αυτό είναι για τους ε, επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Δύο ακόμη επιχειρήσεις, ε, την ε, Αταλάντη στην οποία, για την οποία μίλησα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η οργάνωση της επιχείρησης αυτής η οποία στέφθηκε με τεράστια επιτυχία ε, κινητοποίησε την θαλάσσια βιομηχανία και το σύνολο της ναυτιλίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν πήγα, αν πήγατε στο Northwood, αν είδατε τι έγινε εκεί, θα είδατε ότι υπάρχει μία ε, κοινή διοίκηση στρατιωτική και ε, πολιτική που ε, συγκεντρώνει πάρα πολλούς φορούς, είναι πάρα πολλούς φορείς. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται εδώ και ένα. Είναι όλο και λιγότερη η πειρατεία που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε, τι σχέση θα έχουμε στο μέλλον και άμα μπορούμε ε, να αλλάξουμε το μηχανισμό αν χρειαστεί. Αυτά είναι τα ερωτήματα που τίθενται ε, και η σχέση με την επιχείρηση Σοφία. Ο στόχος είναι, είναι να μεταφραστεί ε, στη, να μεταφραστεί στο να ε, ε, δικαστούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ε, θέτουν σε κίνδυνο τόσους πολλούς ανθρώπους ε, που τους βάζουν μέσα σε καριδότσουφλα, γιατί δεν μπορώ να τις αποκαλέσω βάρκες αυτά τα πράγματα. Υπάρχει και αυτό το, θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την επιχείρηση Σοφία σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Για μένα είναι μάλλον ε, μισογεμάτο το ε, ποτήρι. Έχουν γίνει πολλά καλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Παρατηρητήσαμε ε, μια ύπατη εκπρόσωπο η οποία συμμετείχε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ δυναμική και πάρα πολύ δραστήρια. Μέσα σε τρία χρόνια ήταν τεράστια η πρόοδος υπό την ηγεσία της. Ήταν πραγματικά ε, κάτι πολύ σημαντικό το είδαμε το, στο τέλος του 2013 και αρχές 2004 με την κρίση στην ε, ε, Κεντρική Αφρική, όπως επίσης και με την επιχείρηση στη Μεσόγειο. Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πραγματικά πάρα πολύ αφοσιωμένοι 230.000 ε, στρατιώτες έχουμε όπως είπα η Ιταλία έχει δύο επιχειρήσεις το Ηνωμένο Βασίλειο μία ακόμη η Αυστρία δύο η Γερμανία μία ακόμη ε, η οποία ανέλαβε από την Ισπανία και η Γαλλία βλέπουμε λοιπόν ότι αυτές οι χώρες ηγούνται των επιχειρήσεων αυτών υπάρχει μία εναλλαγή και ότι πολλές χώρες εκπροσωπούνται στην ηγεσία των επιχειρήσεων Υπάρχει και επαφή με ε, το ΝΑΤΟ, είναι πάρα πολύ τακτικές οι συναντήσεις μεταξύ του Γενικού Γραμματέα και της ΥΠΑ της εκπροσώπου. Η σημασία του ενός ή ε, της άλλης ε, στην, στις συνεδριάσεις των Υπουργών Αμήνης αυξάνεται όλο και περισσότερο και το ίδιο ισχύει ε, και ε, σε διεθνές επίπεδο η εξωτερική υπηρεσία ε, δράσης όλο και περισσότερο συμμετέχει και ο κόσμος το γνωρίζει πολύ περισσότερο πλέον. Κάτι ακόμη είναι οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις και εδώ το ποτήρι είναι τουλάχιστον μισογεμάτο 18 χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συμμετείχαν ή συμμετέχουν αυτή τη στιγμή σε επιχειρήσεις μας. Υπήρχαν πάρα πολλοί στρατηγικοί διάλογοι, η Κίνα, η Ιαπωνία, όπως επίσης ε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ε. και όλα αυτά δείχνουν ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικές πρόοδοι, όμως δυστυχώς δεν έχει ξεχυλήσει κιόλα το ποτήρι. Η δυνατότητα ε, ανάπτυξης υποδομών ή κοινέ υποδομές σε ατχό κομμάδες δύο ή τριών ε, είναι σε εμβρυϊκό στάδιο. Ε, έχουμε ακόμη πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες διαδραματίζονται μεμονωμένα από τις χώρες το, η κατανομή του άχθους, του οικονομικού άχθους ε, και, του ανθρώπινου άχθους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, πρέπει να κάνουμε περισσότερο και πρέπει να περισσότερα και να προσπαθήσουμε πολύ περισσότερο. Καταλαβαίνω ο πάντως ότι δεν είμαστε αλλεργικοί στην ανάληψη κινδύνου. Βλέπω ότι στο Μογκαντήσου αναλάβαμε το ρόλο μας με πολύ πιο ε, στεναρό τρόπο και το είδαμε επίσης ε, και στην επιχείρηση που επέτρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, να ε, δραστηριοποιηθούν στην κέντρο Αφρικανική δημοκρατία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό είτε από μικρότερες κλίμακας επιχειρήσεις είτε για τεράστιες κλίμακες επιχειρήσεις. Βλέπω λοιπόν ότι η ανάληψη κινδύνου ε, αλλά δεν ε, είναι, δεν είναι άχρηστη. Ε, γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις στις Βρυξέλλες. Αυτό βέβαια δεν ε, μας απέτρεψε από το να αρχίσουμε τέσσερις καινούργιες επιχειρήσεις και να συνεχίσουμε τις έξι προηγούμενες που είχαμε αρχίσει. Για μένα ε, η Ευρώπη της αλληλεγγύης είναι αυτή που πρέπει να προχωρήσει. Επομένως ε, θεωρώ ότι έχει γίνει γιγάντια πρόοδος κατά τα τελευταία τρία χρόνια και το έχω δει εγώ στο δικό μου ε, περιορισμένο τομέα. Όσον αφορά την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων για κοινά ωφέλη, εκεί είναι τεράστια η πρόοδος που πρέπει να σημειωθεί ακόμη. Πιστεύουμε όλοι ότι βεβαίως αυτό το οποίο ανέλαβε η εκπρόσωπος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν ε, η επεξεργασία νέας στρατηγικής που θα δώσει τη δυνατότητα να εντοπιστεί τι θα κάνουμε σε επίπεδο 28 από κοινού, γιατί αυτή τη στιγμή ε, το εντοπίσουμε, το χτενίσουμε και το καταστήσουμε πιο συγκεκριμένο, θα μπορέσουμε να αναδιοργανωθούμε, θα μπορέσουμε να δούμε ποιοι είναι οι τομείς ε, εμπειρογνωμοσύνης μας, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις κρίσεις μερικές φορές ε, μεμονωμένα, μερικές φορές στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και μερικές φορές επίπεδο 28 σε επίπεδο Ένωση. Αυτά κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, στρατηγέ. Είναι ίσως όντως η τελευταία φορά που βλέπουμε τον ε, στρατηγό υπό την τωρινή του ιδιότητα εδώ στην Επιτροπή μας. Σίγουρα ευχαρίστως θα συναντήσουμε και τον διαδοχό σας αργότερα. πάση περιπτώσει. Τώρα αφού σας ευχαριστήσω συζήτηση. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, στρατηγέ, για την έκθεσή σας. Συγχαρητήρια από τη δική μου πλευρά για τη δουλειά που έχετε κάνει και εύχομαι κάθε επιτυχία και στη συνέχεια. Όπως και εσείς, είμαι και εγώ αισιόδοξο. Έχουμε προχωρήσει, πιστεύω, κατά τα τρία τελευταία χρόνια, κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Θα ήμουν πολύ απογοητευμένος αν ε, δεν ε, είχαμε αντιδράσει καθόλου στην κατάσταση στις γειτονικές μας χώρες. Ε, πρέπει να αντιδρούμε και να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις που προκύπτουν. Συμφωνώ ότι το ποτήρι είναι μισογεμάτο, τελείως γεμάτο όμως δεν είναι και όλα. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε αυτά που εκκρεμούν ακόμα. Αναφερθήκατε στην ε, νέα κοινή πολιτική ασφάλειας ε, και άμυνας που θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τον επόμενο Ιούνιο. Ελπίζω ότι και ο διάδοχός σας θα συνεχίσει να προωθεί τα θέματα αυτά και ότι θα μπορούμε να μιλάμε για συνέχεια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής ε, του 2003 και να μην μιλάμε πολύ γενικά για την ε, μεγάλη αυτή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας και θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν εγκαίρως ώστε να συζητηθεί αναλυτικά αυτός ο τομέας. Αναφερθήκατε και σε έναν άλλον τομέα, command and control. Δεν έχουμε μια ενιαία έδρα, υπάρχει ένα κέντρο ελέγχου μόνο. Τα κράτη-μέλη που πάντα είναι επιφυλακτικά πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Και βλέπω ότι όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, όπως το πρόγραμμα Σοφία, θα πρέπει να τα ελέγξουμε από εδώ, διότι δεν ξέρουμε και πόσο καιρό θα κρατήσουν. Ειδικά για το πρόγραμμα Σοφία. Νομίζω ότι χρειάζεται ε, ο δέον προγραμματισμός για την ε, τρίτη περίοδο. Από πότε θα μπορέσουμε με μια σχετική δομή στη Λιβύη να υπολογίζουμε ότι θα έχουμε συνομιλητές ε, και όσον αφορά την ασφάλεια και όσον αφορά τους μετανάστες, ε, τους πρόσφυγες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σέλερ, παρακαλώ. Πριν αποχωρήσετε, να σας κάνουμε και ένα δωράκι όσον αφορά το σύστημα ελέγχου του Command and Control. Μας είχατε πει ποια είναι τα βασικά εμπόδια. Μπορεί να μην υπάρχει πολιτική απόφαση, αλλά τεχνικά με το, από τον προϋπολογισμό καταφέραμε από τον Σεπτέμβριο να γίνει η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων και Πιστεύουμε ότι μέσα σε τρία χρόνια ε, να μπορέσουμε με ε, δημόσια σύμβαση να χρηματοδοτήσουμε το πρόγραμμα αυτό. Υπήρξαν λοιπόν κάποιες ε, ενέργειες εντός του Κοινοβουλίου και έτσι καταφέραμε να έχουμε αυτή τη γραμμή στον προϋπολογισμό. Η ερώτησή μου έχει και αυτή να κάνει με το Σοφία πέρση, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Είχαμε την απόφαση 2240 που αναφέρεται στις θάλασσες της Λιβύης και πριν από αυτό είχαμε ε, μια απόφαση για τη δημιουργία μιας ε, κυβέρνησης ενότητας ε, στη Λιβύη όπου καλούνταν οι ενδιαφερόμενοι να συνεργαστούν κλπ. Όσον αφορά λοιπόν την εντολή του Σοφία, και λαμβάνοντας υπόψη την αστάθεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Λιβύη, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά σκάφη βρίσκονται ακόμα ε, υπό τον έλεγχο των ε, διαφόρων ε, ενοπλών ομάδων. Υπάρχει λοιπόν πρόγραμμα για να καταστραφούν τα σκάφη αυτά και αν ναι, Πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα Σοφία να αντιμετωπίσει ε, το θέμα αυτό και τον αντίκτυπό του. Άλλη ερώτηση. Πώς επηρεάζει το Σοφία επιχειρήσεις της Frontex όπως είναι η Τρίτον, διότι μπορεί να γίνουν πιο σημαντικές για όλους αυτές οι επιχειρήσεις έχει ληφθεί απόφαση όσον αφορά τη μετάβαση από τη φάση 2 στην φάση 3 από ε, την ε, ε, Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας και όσον αφορά την επιχειρησιακή εντολή, το να αντιμετωπίσουμε μόνο τους διακινητές αφήνει εκρεμές το θέμα των μεταναστών και των ε, μεταναστευτικών οδών. Μου φαίνεται ότι η επιχειρησιακή εντολή είναι μάλλον στενή. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να αναπτύξετε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Έλερο Μάρο Κιούρεκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον στρατηγό. Όπως και οι προλαλήσαντες, ε, χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ στην Επιτροπή μας ε, και μπορείτε να μας μεταφέρετε πληροφορίες που είναι πάρα πολύ χρήσιμες για μας. Έχω μία συγκεκριμένη ερώτηση που έχει να κάνει με το σημαντικότερο επίπεδο στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής άμυνας. Είναι σημαντικό αυτό που οι Γάλλια ε, ονομάζουν πρεζόν, στην παρουσία μας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε σχετική απόφαση και θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η δική σας άποψη, πώς βλέπετε το μέλλον της επιχείρησης αυτής. Εμένα με ενδιαφέρει για τον εξής λόγο. Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της προηγούμενης εβδομάδας έχει να κάνει με το τελικό αποτέλεσμα, αλλά αντιμετωπίζουμε όλο και μεγαλύτερες απειλές, τις οποίες θα πρέπει τουλάχιστον θεωρητικά να εξετάσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι η γνώμη σας, στρατηγέ. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει στη Μεσόγειο. Και έχουμε μια εντολή η οποία αφορά όμως μόνο το ένα μέρος της, ε, το δυτικό μέρος. Ε, τι ισχύει όμως για τους διακινητές στην Μαύρη Θάλασσα. Τα θέματα αυτά θα επηρεάσουν ε, την ασφάλεια των κρατών μελών. Η... Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε νεοεμφανιζόμενες απειλές. Θα υπάρξει εντολή για κινητοποίηση και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Τουρκία που σχετικά με άλλες χώρες είναι πάρα πολύ... Ε, όπου σε αντίθεση με άλλες χώρες είναι πάρα πολύ σταθερή η κατάσταση. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους μας για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Δεδομένης της μαζικής λαθρεπορίας ανθρώπων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Στρατηγέ, λυπούμε πολύ που δεν μπόρεσα να ακούσω τα εισαγωγικά σας ε, σχόλια. Δεν θέλω όμως να χάσω την ευκαιρία να σας ε, κάνω ερωτήσεις. Είχε έρθει η κυρία Μογκερίνη στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ε, και τη ρώτησα για την έλλειψη συντονισμού των κρατών μελών που επιχειρούν στο Ιράκ ε, στην πρώτη γραμμή κατά του ISIS. Πήγα τον προηγούμενο μήνα 10 χιλιόμετρα από τη Μοσούλ, 1,5 χιλιόμετρο από το, την πρώτη γραμμή με τους Πεσμεργά και το ISIS, ε, πραγματικά μου έκανε τεράστια εντύπωση η πολύ ο πολύ ε, κακός εξοπλισμός, παρά το γεγονός ότι ήταν πάρα πολύ γενναίοι, δεν έχω καμία αμφιβολία. Κάποια κράτη-μέλη έχουν πάρα πολύ καλό ε, στρατιωτικό εξοπλισμό λόγω της Γερμανίας που εφοδίασε με, με τάγκς κλπ. Αλλά φυσικά δεν αρκεί για να καλύψει την πρώτη γραμμή που είναι 150 χιλιόμετρα. Δεν έχουν ε, αισθητήρε νυχτό, δεν έχουν πυρομαχικά, δεν έχουν πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι σε μερικές περιπτώσεις η τεχνική δημοκρατία ε, προμήθευσε κάποιο εξοπλισμό. Δεν χρειαζόμαστε ε, περισσότερες, ε, περισσότερα στρατεύματα. Χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό και καλύτερη εκπαίδευση. Τα κράτη-μέλη μας δεν έχουν επαρκή συντονισμό. Η κυρία Μουγκερίνη λέει ότι στο πλαίσιο ε, ε, ε, της συμμαχίας το κάνουν αυτό. Όμως για ποιο λόγο υπάρχει η ΚΕΠΑ αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερο συντονισμός. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, τα κράτη-μέλη δεν καταπολεμούν σωστά το ISIS και φυσικά δεν ανταποκρινόμαστε και στις προσδοκίες των πολιτών μας γιατί δημιουργούμε όλο και περισσότερους πρόσφυγες και δημιουργούμε όλο περισσότερα προβλήματα και εμείς δεν ανταποκρινόμαστε στι προσδοκίε των πολιτών μας ε, κα, κατ' επέκταση. Θα ήθελα να κάνω και μία ερώτηση σχετικά με την επιχείρηση Σοφία. Αφορά μόνο ε, τη θάλασσα ή πηγαίνει πέρα από το θαλάσσιο κομμάτι και επεκτείνεται και το χερσαίο κομμάτι, μήπως ε, συμπεριλαμβάνει για παράδειγμα και ε, αεροπορικές δυνάμεις κλπ. Εντάξει, ε, συμφωνούμε ότι καλό είναι να συνεχίσει αυτή η επιχείρηση, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Ακούσαμε ότι υπήρξε υποστήριξη ε, ε, από την ε, κυβέρνηση. Βέβαια είναι γεγονός ότι υπάρχει κάποια υποστήριξη από τη Σαουδική Αραβία και από τα Εμμυράτα έχουν σκοπό να κάνουν μια επίθεση στην Ιεμένη, κάτι το οποίο θα είναι απολύτως καταστροφικό όσο καταστροφική ήταν και η ρωσική επίθεση στη Συρία. Και γνωρίζουμε ότι η προμήθεια όπλων από την Τουρκία φτάνουν στη Μισράτα και ε, υπάρχει ε, πρόσβαση μετά από τη Μισράτα στην Τρίπολη. Οπότε πώς ε, πώς θα πάει η επιχείρησή μας, πώς θα, πώς κινηθεί αν υπάρξει ακόμη βιαιότερη κατάσταση και εκφυλισμός της κατάστασης ε, στην ε, ε, Συρία. Ευχαριστώ. Thank you, madam. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Αλσακάμ. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον στρατηγό. Εγώ θέλω να μιλήσω για την ασφάλεια. Ξέρουμε τι επιπτώσεις έχει και στρατιωτικά και μη στρατιωτικά. Έχουμε τις κατευθυντήριες γραμμές του 2012. Τι πρόοδο έχουμε πετύχει. Ευχαριστούμε. Κύριε Κάλλερ, έχετε μια ακόμα ερώτηση. Ναι, κάτι ξέχασα που ρωτάω κάθε φορά όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό είναι γιατί δεν προχωράει η μεταρρύθμιση του μηχανισμού Αθήνα. Η χρηματοδότηση είναι πολύ βασικό το κόστος για τις χώρες μέλη προκειμένου να συμμετέχουν περισσότερες. Οπότε θέλω να ξέρω γιατί δεν προχωράμε σε αυτό. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για τις τελευταίες συζητήσεις, αν υπάρχουν βέβαια. Ωραία, δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, λέει η Πρόεδρος. Οπότε και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, επιτρέψτε μου. Διάφορες, αλλά τέλος πάντων κάποιες. Στρατηγέ, μπορείτε να μας πείτε που βρίσκεται ο διάλογος με τις Ηνωμένε Πολιτείες και κατά πόσο στην εμερήσια διάταξη του διαλόγου με την Κίνα περιλαμβάνεται και ο κυβερνοχώρος τι συζητήσει γίνονται από αυτού με την Κίνα. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο, στρατηγέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα αρχίσω με αυτή την τελευταία ερώτηση όσον αφορά τον κυβερνοχώρο. Ναι, λοιπόν, έχουμε τέτοιο διάλογο με την Κίνα, στο Πεκίνο μάλιστα πριν από λίγους μήνες. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να έχουμε σχέσεις με την Ασία, όχι γιατί στρατιωτικά σκοπεύουμε να έχουμε δράσεις εκεί, αλλά γιατί υπάρχουν θέματα για τα οποία θέλουμε να έχουμε συζητήσεις υψηλού επίπεδου. Και αυτό ακριβώς ανέλαβα να κάνω εκεί. Δεν ασχολήθηκα με το, για τον κυβερνοχώρο, με την Κίνα, είναι δηλαδή θέλω να πω πιο πολύ πολιτικό αυτό το ζήτημα. Επικεντρώθηκα όμως στην Αφρική και αυτό γιατί βλέπω ότι η Κίνα εμπλέκεται θετικά βέβαια στην Αφρικανική Ήπειρο. Και το στρατηγείο του Μαλή ε, βρέθηκε με το στρατηγείο το κινέζικο στο Μαλή υπό τον ΟΗΕ τέτοιου είδους επαφές πρέπει να υπάρχουν. Ήμουνα στο Μογκαντήσου πρόσφατα στο αεροδρόμιο υπήρχαν Κινέζοι στρατιώτες. Είναι σημαντικό δηλαδή να κάνουμε τέτοιες επαφές. Τώρα, εκτός Κίνας τώρα, τι πρόοδος έχει γίνει όσον αφορά τον κυβερνοχώρο τα τελευταία χρόνια. Έχει γίνει, αλλά μένουν πολλά ακόμα να γίνουν. Και μερικά δεν θα μπορέσουμε να τα κάνουμε και θα αρχίσουμε αυτά. Ο κυβερνοχώρος είναι απόρριτη υπόθεση, ιδιαίτερα ευαίσθητη και είναι πάρα πολύ δύσκολο να συζητήσει κανείς με περισσότερο από έναν ή δύο. Με 28, όπως καταλαβαίνετε, αποκλείεται. Εμείς και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ασχολιόμαστε με την συνδυτοποίηση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Συνειδητοποίηση των απειλών που υπάρχουν στον κυβερνοχώρο. Τέτοια θέματα συζητάμε. Αλλά υπάρχει και κάτι στο οποίο δεν έχουμε κάνει πρόοδο καθόλου. Και αυτό είναι βέβαια πιο πολιτική συζήτηση από αυτού, δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Είναι και τις χώρες που δεν έχουμε δράση σκέπα. ...που δεν υπάρχει στρατιωτική στήριξη. Υπάρχει μια ρήτρα αλληλεγγύης με τα τελευταία γεγονότα είτε για τη μετανάστευση είτε για άλλα χρησιμοποιούνται στρατιωτικές δυνάμεις που δεν είναι δράση και έπα. Ξέρουμε ποιες είναι οι συνέπειες του κυβερνοχώρου. Κάποια στιγμή, κάποια χώρα θα έχει ξεπεραστεί και δεν θα μπορέσει από μόνη της να λύσει τα ζητήματα. Και γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε όλοι εδώ στις Βρυξέλλες ότι οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό, τον κυβερνοχώρο, είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να προχωρήσουμε. Εμείς κάνουμε το σχεδιασμό, ε, ξέρουμε τι εργαλεία μπορούμε να προσφέρουμε, πέρα δηλαδή από την στρατιωτική πτυχή. Μένουν πολλά να γίνουν, αλλά έχουν γίνει και πολλά. Κύριε Γκόμες, θέλω να επιστρέψω στο πρώτο τμήμα της ερώτησής σας, που είχε να κάνει με το Ιράκ, τη Μοσούλ. Ήμουνα πριν από χρόνια και για την επέκταση του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους και πώς οι διάφορες χώρες μέλη επιδρούν στα θέματα του εξοπλισμού και της εκπαίδευσης. Δεν μπορώ να σας απαντήσω για τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και το ξέρει η Επιτροπή σας και το ξαναλέω, ότι μία από τις πιο αποτελεσματικές μας δράσεις από πλευράς Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σομαλία με τις αμυντικές αρχές αργότερα και στην Κεντρική Αφρική. Και είναι το θέμα του εξοπλισμού. Γιατί δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού εξοπλισμό. Οι χώρες μέλη δεν θέλουν να κάνουν περισσότερα από αυτά που ήδη κάνουν ε, μέσω των σταθιωτικών τους υποχρεώσεων σε αυτές τις χώρες και δεν θέλουν να χρηματοδοτήσουν επιπλέον. Οπότε γι' αυτό και η εταιρική σχέση έχει μεγάλη σημασία. Πολλές φορές με τερική σχέση μπορούμε να βρούμε κονδύλια. Πάντως, εξοπλισμός κατάρτιση σίγουρα είναι κάτι πολύ σημαντικό και εξετάζεται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Πράγματι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό, να έχουμε πρόοδο, να μην παίρνουμε μόνο πολιτικές αποφάσεις, να μην έχουμε προσδοκίες από τις χώρες μέλη και μετά να μην υπάρχουν οι δυνατότητες. Για τον κύριο Γκάλερ, στην ερώτησή σας για το που βρισκόμαστε στο command and control. Αν θέλουμε αυτονομία εδώ στις Βρυξέλλες, πρέπει να χτίσουμε το θέλουμε? Όχι. Σε μερικές περιοχές όμως, σε όλες τις αποστολές κατάρτισης, θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να επιβλέπουμε αν μη τι άλλο αυτές τις δράσεις, τις επιχειρήσεις. Είναι μια συνολική προσέγγιση. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλα τα στοιχεία. Τι γίνεται δηλαδή μέσα στη χώρα, κατάρτιση και εκτός, όπου και ΕΚΟ, ΔΡΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεπώς, το C2 είναι μη εκτελεστική δράση, πολύ χρήσιμη. Αλλιώς, κάποιοι ξέρετε για την Αταλάντα πήγατε. Είναι διαφορετικά τα πράγματα στην πραγματικότητα από ό,τι φαίνονται από τη Ρώμη. Δεν είναι καθαρά στρατιωτικό το θέμα, όπως ε, στον Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας τη Europol, τη Eurojust, διάφορους εταίρους στην περιοχή όχι όμως με τον ναυτιλιακό κλάδο. Το ΝΑΤΟ έχει μια επιχείρηση και όλοι αυτοί οι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οπότε για να απαντήσω για το C του, ναι, υπάρχει θέμα και το κύριο είναι ότι είναι στον σχεδιασμό των ικανοτήτων μας γιατί δεν έχουμε αρκετές ικανότητες. χρειάζονται όλο και περισσότερο εκείνοι οι οποίοι μπορούν να αναλύσουν και να συμβουλεύσουν. Όταν έχετε πολλούς πυράβλους από την Κασπία πάνω από το Αφγανιστάν, Ιράκ, Ιράν, Συρία ίσως, τότε πρέπει να έχετε κάποιον ο οποίος είναι σε θέση να αναλύσει το τι συμβαίνει. Και γι' αυτό εδώ στις Βρυξέλλες χρειαζόμαστε αυτήν ακριβώς την ικανότητα αξιολόγησης και σχεδιασμού. Για το μηχανισμό Αθήνα. Στην αρχή αναφέρθηκα, ελάχιστη πρόοδος έχει γίνει. Είναι θέμα χωρών μελών. Οι χώρες μέλη δεν θέλουνε. Υπάρχει όμως ένας τομέας το u Battle Group. Έχουμε επιχειρήσεις που δεν είναι στρατιωτικές, όπως το NRF, στην Τουρκία, που είναι η ανακούφιση από καταστροφές. Εδώ υπάρχει ενισχυμένη κοινή χρηματοδότηση που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική. Και η Ισπανία που συμμετείχε έχει κακές εμπειρίες. Τους κόστησε πολλά χρήματα ενώ κανένας άλλος δεν βοήθησε. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να πιέζουμε μήπως υπάρχουν το όπου ο μηχανισμός αυτός Αθήνα να μπορεί να βοηθήσει να μοιραστούμε το βάρος. Το είδαμε και με την κρίση του ιού έμπολα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε μεταφορά ασθενών Οπότε και εκεί υπάρχουν τομείς συνεργασίας, θέλω να πω. Έρχομαι τώρα στην Σοφία, που είναι 13 σημεία. Όπως και με την Αταλάντα, από την αρχή ξέραμε ότι το στρατιωτικό στοιχείο ήταν ένα μεταξύ άλλων. Και ξέρουμε επίσης ότι πρέπει να εμπνευστούμε από αυτό που έκανε η Ισπανία πριν από πολλά χρόνια. Έχει να κάνει με τις χώρες προέλευσης πρώτα απ' όλα, σχέση μαζί τους, με τις κοινότητες, με την κυβέρνηση, αναπτυξιακή βοήθεια. Πολλά μπορούν να γίνουν ε, εκεί. Συνεργασία επίσης με τις χώρες transit για να ε, διώκονται και να καταλήγουν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο ζήτημα και υπάρχει και το θέμα στη θάλασσα. Και όπως είπα και στην αρχή, η επιχείρηση αυτή είναι για να σώζονται ζωές. Για να αποφεύγεται ο κόσμος να μπαίνει σε υπερφορτωμένα ερήπια σκάφη χωρίς καύσιμα καλά-καλά που κινδυνεύουν να βουλιάξουν ανα πάσα στιγμή. Και δεν πρόκειται μόνο για στρατιωτικές φρεγάτες και άλλα πλοία, υπάρχουν και υποβρύχια και άλλος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζονται τα σκάφια αυτά. Είναι επιχειρήσεις για να σώζονται ζωές. Και δεν είναι δευτερεύον, είναι κεντρικό. Η επιχείρηση Σόφια δηλαδή έχει σώσει χιλιάδες ζωές πρόσφατα. Πάντως, όπως είπαμε και στην αρχή, στόχος είναι να δείξουμε με όλα τα μέσα και με πλήρη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και με τη Συμφωνία της Λιβύης, να πηγαίνουμε εκεί που χρειάζεται για να καταστρέφουμε αν χρειάζεται που σημαίνει και, στη, και αν χρειάζεται, εφόσον χρειάζεται και εφόσον μας το έχουν ζητήσει. Συνεπώς, ναι υπάρχει σχεδιασμός αλλά είναι ένας αρχικός σχεδιασμός που συμπεριλαμβάνει συγκέντρωση πληροφοριών και ανάλυση και που γίνεται στο στρατηγείο μας. Και από εκεί και πέρα σε καθημερινή βάση συνεργαζόμαστε με τη Europol και την Eurojust. Συμμετέχουν και εκείνοι στο στρατηγείο μας και εμείς πηγαίνουμε εκεί σε συνεργασία με την Τινησία, με την Αίγυπτο γιατί μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο στόχος δεν είναι η χρήση στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά η συγκέντρωση πληροφοριών για να δούμε ποιος είναι ο πιο κατάλληλος για να ανταποκριθεί. Είτε πρόκειται για συνεργασία χωρών, είτε πρόκειται για την ε, μελλοντική προσωρινή κυβέρνηση. Είναι πολλές οι δυνατότητες. Η μετάβαση τώρα από το ένα στάδιο στο άλλο είναι μια πολιτική διαδικασία. Η δράση μας είναι στα ανοιχτά της θάλασσας αποκλειστικά και από εκεί να περάσουμε στα χώρια ύδατα αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση από το Συμβούλιο που, σημαίνει ότι αν Λεκράν θα μου γράψει, θα το δει η Επιτροπή μας, θα το δει επίση, μετά θα γίνει η αξιολόγηση, το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει ότι ναι, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο και μετά οι πρέσβες του πίση, θα αποφασίσουν το πότε θα γίνει αυτό. Κάθε ένα από αυτά τα στάδια είναι πολύ συγκεκριμένο και προδιαγραμμένο πολιτικά για προφανείς λόγους, γιατί αλλάζουν οι σχέσεις σε διεθνές επίπεδο, οπότε δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από μια στιγμή στην άλλη. Ο Άμιλ Κρέιν γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να εφαρμόσει το ίδιος μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε, που είναι ο μηχανισμός που σημαίνει ότι υπάρχει δράση και αντίδραση που λαμβάνει υπόψη όλους τους εταίρους. Και οι εταίροι αυτοί είναι διάφοροι παράγοντες που δρούν γύρω από τη Λιβύη. Και νομίζω ότι έτσι απάντησα, νομίζω, στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Στρατηγέ, θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι ο Ναύαρχος Κρέτιντίνο της UNAFOR ε, ε, ε, Σοφία θα έρθει στη, την 1η Δεκεμβρίου και θα έχετε τη δυνατότητα να συζητήσετε μαζί του τις διάφορες λεπτομέρειες της γνωστής αυτής πλέον επιχείρησης. Θα ήθελα τώρα να σας ε, ε, να ευχαριστήσω τον ε, στρατηγό για την υπομονή του, για την καλοσύνη του να είναι εδώ μαζί μας σήμερα, ώστε να ενημερώσει την υποεπιτροπή μας για τις εξελίξεις στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, όπως επίσης και τις διάφορες αποστολές κάθε φορά που του ζητούμε να παραστεί στην Επιτροπή μας είναι πάρα πολύ πρόθυμος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλη μου χαρά, λέει ο στρατηγός.